Okay. Um, λοιπόν, θα αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση που θα συνεχιστεί αύριο το απόγευμα, όπως θυμόσαστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Φαίνεται ότι ναι. Σημείο 2. Τα πρακτικά συνεδρίαση 23 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. υπάρχουν στο φάκελό σα. Εάν μέχρι το τέλος της ημερησίας διάταξης σήμερα δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, για τα πρακτικά θα θεωρήσουμε ότι αυτά έχουν εγκριθεί. Σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Ανακοινώσει Προέδρου. Θα ήθελα να σας πω στο σύνολο ότι έχουμε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού στη Σοκχόλμη που πήγε τον Δεκέμβριο συναντήσαμε τέσσερους είδους ε, υπουργού που καλύπτουν διάφορε τομείς της αρμοδιότητάς μας. Και συζητήσαμε τα αποτελέσματα της Σουηδικής Προεδρίας. Επίσης, συζητήσαμε διάφορους εκπροσώπους πανεπιστημίων και καθηγητές για την διαδικασία της Μπολόνια, την πολιτική για την Ούλια και την επικοινωνία. Πήγαμε επίση και στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεργάζονται παραδειγματικά στη Στοκχόλμη. Θέλω να το τονίσω, δεν συμβαίνει αυτό παντού, αλλά στη Στοκχόλμη ναι. Είχαμε και την ευκαιρία να συναντήσουμε διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Καθώς επίσης συζητήσαμε την Υπουργό που είναι αρμόδια για την ασωμάτωση των μεταναστών. Επίσης επισκεφτήκαμε δύο πολιτιστικά προγράμματα, το Θαυμάσιο Σύγχρονο Μουσείο και ένα μουσείο που παρουσιάζει την ε, πολιτική γενικά και τον πολιτισμό των Σουηδών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κύριους Κρίστη Πάκελα και ο Φτάσης που μας συνόδευσαν. Έχετε στα, στο φακελό σας επίσης την έκθεση της αντιπροσωπείας αυτής. Σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χαιρετήσω εγκαδιότατα τον Ισπανό Υπουργό Παιδείας, Ανχέλ Καμπιλόνο, που εκπροσωπεί προφανώς την Ισπανική Προεδρία, και θα ήθελα να χαιρετήσω μέσα και όλους τους Ισπανούς από ό,τι βλέπω που υπάρχουν στην αίθουσα. Σας χαιρετίζω και σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και το Συμβούλιο των Υπουργών είναι εταίροι. Ε, πολλές φορές δεν αγαπούν αλλήλους και πολλοί, αλλά προσπαθούν να συνεργαστούν. Γιατί και οι ΜΕΝ και η ΔΕ έχουμε κατά νου να εξυπηρετήσουμε το οφελό των πολιτών. Και για οποιαδήποτε πρωτοβουλία εξαρτώμεθα η ΜΕΝ από τους ΔΕ. Γι' αυτό καλούσαμε πάντα του υπουργού που ήρθαν πολύ ευχαρίστω. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τον Υπουργό Παιδεία. Αύριο θα συναντήσουμε τον Υπουργό Πολιτισμού. Από ό,τι κατάλαβα, οι προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία είναι καταρχήν ο εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων που συζητήσεται στενά με διαδικασία τη Μπολόνια και μετά ε, το θέμα τη κοινωνική διάσταση τη παιδεία. Οι προτεραιότητες αυτές συμφωνούν με αυτά που συζητάμε και εμείς εδώ αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Ο συνάδελφος Κάρου Σμιτ που είναι και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που έργαζε, προετοιμάζει μια έκθεση για το University Business Dialogue και η κυρία Μαρία Κούτσικ προετοιμάζει μια έκθεση για το θέμα Education and Training, ε, παιδεία και ε, κατάρτιση 2010. Συζητάμε και για την Πολόνια. Δεν είμαστε βέβαια εμεί αρμόδιοι. Είναι τα κράτη-μέλη αρμόδια και τα πανεπιστήμια. Δεν τα έχουν κάνει πολύ καλά τα πράγματα όπως τα έπρεπε, αλλά ελπίζω ότι εσείς ε, θα μπορέσετε κάτι να προωθήσετε με τη συνεργασία της Κομισιόν και των άλλων Υπουργών. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα για 15 λεπτά να πάρετε το λόγο και να μας παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να σας υποβάλουμε ερωτήσεις. Και ελπίζω ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία να σας υποβάλουμε πολλές ερωτήσεις. Γιατί χρειάζομαι καλές απαντήσεις και καλούς εταίρους, όχι αντιπάλους από τη μεριά του, Υπουργού, του, Υπουργείου, του Συμβουλίου Υπουργών. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξότιμοι κύριοι, εμφανίζομαι για πρώτη φορά εν ώψη τη Επιτροπή Παιδεία και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σα παρουσιάσω του στόχου ε, τη Ισπανική Προεδρία ε, στο θέμα τη ε, παιδεία. Η παιδεία φέρει τι ευρωπαϊκέ αξίε τη ισότητα και ο στόχο τη Ισπανική Προεδρία θα είναι να έχουμε περισσότερη παιδεία ποιότητα και για όλου παιδεία δεν αποτελεί τμήμα των μεγαλών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όπως ξέρετε δεν έχει κυρίαρχο χαρακτήρα η εκπαίδευση στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά ε, παρόλα αυτά η Ισπανική Προεδρία θα θέσει τις εκπαιδευτικές αξίες αν οποιοδήποτε ε, συζήτηση σε πιο διορθωτικού χαρακτήρα, πρατώντας αυτό συνεισφέρουμε στο να οικοδομήσουμε την Ευρώπη της γνώσης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα θα συνεισφέρουμε τα μάλλα στην ίδια διαδικασία κατασκευής και ολοκλήρωσης μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ότι το έργο που θα αναπτύξουμε απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνένεση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά δεν μπορούμε ε, παρά να είμαστε φιλόδοξοι στις προτάσεις μας για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Είναι ουσιαστική η στήριξη των ομάδων αυτού του Κοινοβουλίου, που όχι μόνο εκπροσωπούν όλους τους πολίτες ε, των χωρών που αποτελούν την Ένωση, αλλά έχουν και έναν ενισχυμένο ρόλο τώρα με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνα. Θέλω να πω ότι Επίση, χρειαζόμαστε και τις δικέ σας προτάσεις και τις δικέ σας πρωτοβουλίε για να μετοποιήσουμε τις προκλήσεις της εκπαίδευση στο μέλλον. Και σε αυτό το κοινοβούλιο αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ε, θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, της Ισπανικής Προεδρίας ε, για το θέμα της παιδείας, όμως βρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και έτσι είναι περισσότερο απαραίτητο σήμερα η όθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης σε πιο βιώσιμο στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος της Ισπανικής Προεδρίας αυτό το εξάμενο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση με την πεποίθηση ότι είναι δυνατή μια νέα οικονομία στην υπηρεσία του, της κοινωνικής ευημερίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε ένα νέο ε, οικονομικό μοντέλο που να βασίζεται στην εκπαίδευση, στη γνώση, στην καινοτομία και στη διαβίωση στην κοινωνία. Ξεκινώντας από αυτές τις γενικές σκέψεις, οι προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι εξή. Να θέσουμε την παιδεία στην καρδιά της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Δεύτερο, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης. Τρίτο, να προωθήσουμε τις δεξιότητες, τις βασικές δεξιότητες προς στήριξη των νέων ικανοτήτων για ε, ε, θέσει εργασία, να προωθήσουμε τέταρτον τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Γνώσης ως σύγκληση των δύο μεγάλων χώρων υποκοδόμηση στην Ευρώπη, του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεσκαλίας, στην Ανώτερη Εκπαίδευση και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας εξυγχρονίζοντας και ε, καθιστώντα διεθνή τα πανεπιστήμια μας. Αυτές οι γενικές γραμμές ανταποκρίνονται στην ευούληση να ενισχύσουμε την ιδέα μια κοινωνική Ευρώπης μέσω ενό νέου δεσμού μεταξύ οικονομία και παιδεία. Να θέσουμε την παιδεία, την εκπαίδευση στο κέντρο τη οικονομία. Γι' αυτό εργαστήκαμε, εργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Σουηδική Προεδρία και το Τρίο των Προεδριών στην ανάπτυξη, στην κατάρτιση μια πολιτική στρατηγική, έτσι ώστε τα δύο ε, επίσημα συμβούλια παιδεία που θα λάβουν χώρα 15 Φεβρουαρίου στι Βρυξέλλε και 10 και 11 Μαΐου επισκεπτήσει στι Βρυξέλλε να υιοθετήσουν καθοριστικά συμπεράσματα για τη βελτίωση τη ε, εκπαίδευση ε, στι πτυχέ αυτέ. Είμαι πεπισμένο ε, ότι συμμερίζεστε μαζί μου αυτέ τι αρχέ δράση και ότι η Ευρωπαϊκή πολίτες που εκπροσωπείται και τα κράτη-μέλη συμφωνούν στην αναγκαιότητα να τεθεί η παιδεία στο κέντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα έτη αν ε, πρόκειται για το να θέσουμε την εκπαίδευση στην στρατηγική για το 2020, η Ισπανική Προεδρία θα εργαστεί επί των τέσσερων στόχων που συμφωνήθηκαν στο στρατηγικό πλαίσιο για την παιδεία να θέλουμε να καταστήσουμε πραγματικότητα τη διαβίου μάθηση και την γεννητικότητα. Δεύτερον, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Τρίτον, να προωθήσουμε την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Τέταρτον, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα σε όλα τα επίπεδα τη εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, η κοινή εργασία των κρατών μελών και της Κομισιόν θα βασιστεί στην ενίσχυση της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού με επιλογή στοχών δικτών των αμοιβαίων μάθηση ανταλλαγή και επιλογής ε, καλύτερων και νέων πρακτικών. Σε σχέση με τη διαβίου μάθηση ε, θα εργαστούμε στην προσαρμογή των αποτελεσμάτων και ε, την αξιολόγηση της μάθησης και μάλλον των προσόντων της μάθηση στι ανάγκε της αγορά εργασία, αλλά θα εργαστούμε και στο να απαντήσουμε στις κοινωνικά αιτήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων και θα έχουμε έχουμε πιο ευέλικτη στάση ε, και θα χρησιμοποιήσουμε την άτυπη και την ανεπίσημη μάθηση. Έτσι λοιπόν θα λάβει χώρα μια διάσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος διαβιομάθησης ε, που θα ξεκινήσει συζήτηση για την δημιουργία νέων προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στις επόμενες προεδρίες. Τέλος, θα εμβαθύνουμε στην αναζήτηση συνεργειών μεταξύ της διαδικασίας της Μπολόνια για την ανώτερη εκπαίδευση της διαδικασία της Κοπενχάγης ε, για την επαγγελματική κατάρτιση το στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία το 2020. Ε, γνωρίζω ότι ε, η επίτευξη των στόχων αυτών ξεπερνά την ε, εκπεριτροπής προεδρία μιας χώρας, αλλά ο δικό μα ορίζοντα δεν πρέπει να είναι το πρώτο εξάμεινο του 2010, αλλά η ευημερία των μελλοντικών γενεών τη Ευρώπη. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η εκπαίδευση. Τίποτα δεν μα εξισώνει περισσότερα από την πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τι συνθήκε αφιτηρίε. Έτσι, λοιπόν, το κοινωνικό θέμα και η ισότητα των ευκαιριών θα είναι προτεραιότητα στη δική μα Προεδρία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το 2010 είναι το ευρωπαϊκό έτο κατά τη ε, ανέχεια και του κοινωνικού υποκλεισμού και η δική μα Προεδρία θα δραματίσει ξεχωριστό ρόλο εκεί. Και να σα πω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο καταπολέμησης του αποκλεισμού παρά η επέκταση και βελτίωση τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση ω ως εγγύηση ε, προσωπικής ανάπτυξης και απασχολησιμότητα. Τα κράτη-μέλη τη Ένωση έχουν ε, πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε κοινέ προκλήσει, όπω να εγγυθούμε την πρόσβαση σε συνθήκε ισότητα, την ε, προσχολική και σχολική εκπαίδευση, την καταπολέμηση τη πρόορη εγκαταλείψη του σχολείου σε όλα τα επίπεδα, τι ε, πολιτικέ ε, τη εκπαίδευση ένταξη για μαθητέ με ειδικέ ανάγκε και η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, όπω οι μετανάστε ή πολιτιστικέ μειονότητε. Γνωρίζουμε ότι ε, το μέλλον απαιτεί πολιτικές ε, πρόσβασης ε, και εξάλληψη των συνόρων έτσι ώστε να έχουν μια ποιοτική εκπαίδευση. Πρέπει να προωθήσουμε την ένταξη και την ποικιλομορφία και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για την ένταξη των ατόπων που έρχονται από άλλε χώρε για να αποφύγουμε κοινωνικέ συγκρούσει και να διασφαλίσουμε την μελλοντική οικονομική και κοινωνική ευημερία έναντι τη προοπτική γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Επίση, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση τη οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου τη ανώτερη εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια έχουν τη διαβίβαση τη γνώση και την ε, έρευνα αλλά και τη δημιουργία τη γνώση αλλά επίσης πρέπει να εγγυώνται την επιστροφή στην ε, κοινωνία μέσω της καινοτομίας και της διαβίβασης του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων τους και μέσω υποτροφιών ε, και ε, άλλων, άλλου τύπου βοήθειας πρέπει να καταστήσουμε ρεαλιστική αυτή τη διαβίβαση. Έτσι λοιπόν η Ισπανική Προεδρία θα οργανώσει τι επόμενε διασκέψει. 11 και 12 Μαρτίου θα γαλεύει χώρα στη Μαδρίτη η συνδιάσκεψη, η εκπαίδευση τη ε, ένταξη, οδό για να ευνοηθεί κοινωνική συνοχή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ειδικών ε, ε, εκπαιδευτικών αναγκαιοτήτων. Στις 27 και 28 Μαΐου στην Μάλαγα θα λάβει χώρα η συνάντηση με τίτλο «Διάσταση και κοινωνική ευθύνη των πανεπιστημίων». Κυρίε και κύριοι, ε, θέλουμε να αναπτύξουμε νέες δραστηριότητες. Ε, το 2006 εγκρίθηκε μία σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ε, δραστηριότητες, για τις δεξιότητες κλειδιά, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη διάρκεια όλης της ζωής. Ε, το 2009 τα κράτη-μέλη προτίμασαν εκθέσει για μια πρώτη αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο. Η σύνθεση αυτών των εκθέσεων θα θετηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2010 στο ε, Συμβούλιο Παιδεία. Αυτές οι δεξιότητες ε, πρέπει να αναπτύσσονται κυρίως στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το νέο οικονομικό μοντέλο απαιτεί επαγγελματική κατάρτιση που να προσαρμόζεται στι αναγκαιότητε μια βιώσιμη οικονομία και τη αγορά εργασία, που να ενδυναμώνει του αναδυόμενου τομεί που να εντάσσει την κατάρτιση ε, στου τομεί τη παιδεία και στον επιχειρηματικό τομέα. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίζει και να εντάσσει την επαγγελματική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν και θα ανανεωθούν προτεραιότητε των κοινοτικών πολιτικών ε, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Θέλουμε να προωθήσουμε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματο μονάδων επαγγελματική κατάρτιση και του πλαισίου αναφορά εγγύηση ποιότητα για την επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι, θέλουμε να αυξήσουμε την κινητικότητα και να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε νέε μορφέ μάθηση. Η Ισπανική Προεδρία έχει προβλέψει να οργανώσει στι 5 και 6 Μαου στη Σαραγώσα μια συνδιάσκεψη όπου θα συζητηθούν οι διάφορες διαδικασίες που διευκολύνουν την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της εργασιακής εμπειρίας και των άτυπων τρόπων κατάρτισης ως ε, σημαντικού παράγοντα για τη βελτίωση της πρόσβασης και την προώθηση στην ε, απασχόληση, την προαγωγή στην απασχόληση, όπως και για να διευκολυνθεί η διαβίου μάθηση. Όπως ξέρετε, το 99 τα κύρια ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συναντήθηκαν στην ε, Μπολόνια ε, όπου συμμετείχαν και κάποιοι υπουργοί παιδείας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Το να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος ανώτερης ανάπτυξης σημαίνει ότι Έχουμε ε, ένα μεγάλο σχέδιο εναρμόνιση των ευρωπαϊκών συστημάτων. Όμω δεν ζητούμε εδώ την ε, ομοιομορφία, αλλά ζητάμε την ποικιλομορφία. Τα πανεπιστήμια θέλουμε να έχουν παρόμοια δομή και αυτό ξεπερνά τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, γιατί συμμετέχουν 46 χώρε από όλη την Ήπειρο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συστήματα συγκρίσιμα και συμβατά, όχι απαραίτητα ταυτόσιμα αυτό θα διευκολύνει την κινητικότητα και την ε, αναγνώριση. Η σύγκληση απαιτεί ε, το συντονισμό στις ε, πολιτικές των πανεπιστημίων των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό. Μεγαλύτερη αυτονομία για τα πανεπιστήμια, συστήματα αξιολόγησης απαιτητικού χαρακτήρα, αύξηση και επικοινομορφία των πηγών χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, πιο διαφανής διαχείριση των πανεπιστημίων, μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών μεγαλύτερη ε, ισονομία στο σύστημα και άνοιγμα των πανεπιστημίων στην κοινωνία. Τέλος, ε, αυτή είναι η διαδικασία της Βολονία, να κάνουμε σταθερά βήματα προς την ποιότητα και την αριστεία στο πλαίσιο αυτό της ε, ισονομίας. Θέλουμε μεγαλύτερη ένταξη μεταξύ της ανώτερης εκπαίδευσης και της καινοτομίας και γι' αυτό θα έχουμε στο Σαντιάγο μια συνδιάσκεψη για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο και όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τη ε, Μπολόνια, θα δοθεί περαιτέρω εμβάθυνση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερη Εκπαίδευση και θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ένα νέο ε, πλαίσιο σύμφωνα με την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Γνώση. Ε, η Κομισιόν έχει καταρτήσει μια στρατηγική εξυγχρονισμού των πανεπιστημίων και εμεί θέλουμε να προωθήσουμε την μεταρρύθμιση των μαθημάτων, την κοινωνική ευθύνη του Πανεπιστημίου και την πρόθεση τη έρευνα. Και σε αυτά τα δύο λεπτά που μου μένουν, θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, η κυρία Βιένα Δύο, Υπουργό ε, Ισότητα τη Ισπανία, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα στην Επιτροπή αυτή, γιατί παρευρίσκεται σε μια συνεδρίαση τη ε, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των Διοφύλων και μου ζήτησε εξ ονόματο τη Ισπανική Προεδρία να παρουσιάσω τι προτεραιότητε στον τομέα τη νεολαία. Εγώ θα παρουσιάσω πολύ γενικά τις προτεραιότητες αυτές, γιατί ξέρετε εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός, και επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο δεν μπορώ να αναφερθώ σε βάθος όμως είναι στη διάθεσή σας οι προκοσιότητες για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Τη 1η ε, Ιανουαρίου τέθηκε σε εφαρμογή το ενωμένο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Συνεργασίας για την ΕΟΛΕ για την περίοδο 2010-2018 που εγκρίθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών στις 27 Νοεμβρίου 2009 και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Ένα από τα κύρια ε, μέσα που εισάγει το πλαίσιο είναι ο διαφερωμένο διάλογος μέσω της ενεργής συμμετοχής των νέων στις πολιτικές, των οποίων είναι αποδέκτες για να διασφαλίσουμε τη σωστή ε, παρακολούθηση και λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Σήμερα το πρωί δημιουργήθηκε η ε, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καθοδήγησης. Αυτή η Επιτροπή ε, θα είναι το Φόρουμ Προετοιμασία των Συνδιασκεψίων Νεολαία Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών Προεδριών. Η πρώτη από αυτέ τι συνδιασκέψει με τίτλο Η απασχόληση των νέων ω ε, εργαλείο για την κοινωνική ένταξη θα λάβει χώρα 13 έω 15 Απριλίου στο Χέρι Δελα Φροντέρα στην Κάντι. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεολαία έγγραφο κλειδί στο θέμα αυτό που εντάχθηκε στρατηγική τη Αβώνα θα είναι στο τέλο του. Το να ότι το περιεχόμενό του ε, πέρα από το να διατηρηθεί θα ενισχυθεί και θα προωθηθεί στο νέο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 ε, έχει Πολύ μεγάλη σημασία. Η Ισπανική Προεδρία ε, θέλει να σχεδιάσει ειδικά μέτρα που απευθύνονται ε, στους νέους υπό ε, μέσα από το να δώσουμε νέες ικανότητες στους νέους, κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες η Ισπανική Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών στις 11 Μαΐου θα παρουσιάσει συμπεράσματα για το μέλλον του Συμφώνου της Νεολαίας. Η σημερινή οικονομική κρίση θίγει ιδιαίτερα τους νέους ε, και εξού και η σημασία της εκπαίδευσης και δεδομένου ότι το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η Ισπανική Προεδρία θα παρουσιάσει μια πρόταση ψηφίσματος για την ενεργή ένταξη των νέων και την καταπολέμηση της ανέχειας και της ανεργίας. Κυρίε και κύριοι Πρόεδρο, ε, η Πρόεδρε, κλείνω εδώ. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να απαντήσουν στο αίτημα εκατομμυρίων ε, πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μα ζητούν περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη πρόοδο και περισσότερη ευημερία για να αντιμετωπίσουν ε, τι μελλοντικέ προκλήσει τη Ευρώπη. Γι' αυτό σα επαναλαμβάνω ότι είναι θεμελιώδε να θέσουμε την παιδεία στο κέντρο των κοινοτικών πολιτικών και θα ήθελα να τίνω τη χείρα σε όλες τις κοινοβουλευτικές ε, ομάδες ε, για να εργαστούμε από ε, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βούληση και την επιθυμία επίτευξη συμφωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ισπανική Προεδρία δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην παιδεία. Βεβαίω και εσεί είσαστε Υπουργό Παιδεία και αυτή είναι η αρμοδιότητά σα. Και είμαι σίγουρη ότι όταν πρόκειται για τη δημοσιονομική προοπτική για τα νέα προγράμματα, οποτεδήποτε το συζητήσουμε αυτό, τότε είμαι σίγουρη ότι η Ισπανία θα συμφωνήσει μαζί μας να προβλεφθούν περισσότερα κονδύλια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ζήτησαν πάρα πολύ το λόγο. Ε, παρακαλώ ή δυνατόν να είσαστε σύντομοι, ε, να κάνετε ερωτήσεις και να μην κάνετε τη δική σας την εισήγηση, έτσι ώστε ε, να υπάρχει να υπάρχουν ερωταπαντήσεις. Ο συνάδελφος κύριος Φίσας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την πολύ πλήρη έκθεση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της κινητικότητας, όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και των καθηγητών και όχι ως απλώς προσκεκλημένων καθηγητών, αλλά υπάρχει όπως ξέρετε και το θέμα των διαγωνισμών στη χώρα μας, αλλά και θα ήθελα να αφαιρθώ στη δυνατότητα ε, καθηγητές από πολλές χώρες να μπορούν να διδάσκουν σε άλλα πανεπιστήμια άλλων χωρών. Έχουν προβλεφθεί κάποια μέτρα για να διευκολυνθεί αυτή η δυνατότητα διδασκαλίας ε, σε διαφορετικά ε, πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με το σχάρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωμα οποιοδήποτε εργαζομένου να εργαστεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπετε κάτι τέτοιο για τους καθηγητές. Molte grazie Presidente, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να, να συγχαρώ τον Υπουργό για το σθένος με το οποίο παρουσίασε την εκπαιδευτική πολιτική και πώς έχει τεθεί η πολιτική αυτή στις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας τον επόμενο Μαρτίο στη Βουδαπέστη. Για μια ακόμη φορά θα υπάρχει υπουργική συνδιάσκεψη στα πλαίσια της διαδικασίας της Λισαβόνας ε, για να προετοιμαστούν οι στόχοι του 2020. Η διαδικασία της ε, Μπολόνια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό Σαπατέρο, ε, με πολύ καλές λόγια είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Όμως υπάρχουν δυσκολίες και κυρίως ε, σε κάποιες ε, χώρες ή υπουργικές ε, συνεδριάσεις που καθορίζουν σημαντικούς στόχους δεν κατορθώνουν παρόλα αυτά στα περιφερειακά πανεπιστήμια ούτε φτάνουν στους καθηγητές. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια μέτρα θα υιοθετηθούν για να, για να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότεροι πρωταγωνιστές ε, στη διαδικασία αυτή. Λόγου χάρη το quality assessment ε, του deployment supplement tuning. Αναφέρω συγκεκριμένους στόχους που όμως δεν προχωρούν επαρκώς προκειμένου να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των πανεπιστημίων γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση για να υπάρχει αναγνώριση των πτυχίων από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Τώρα το δεύτερο αφορά την εκπαίδευση. Άκουσα τα λόγια σας ε, και ε, είπατε ότι η εκπαίδευση είναι στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, αυτή η υπεποίθηση πρέπει να ξεπεράσει ένα δισταγμό του Συμβουλίου στο παρελθόν να ασχοληθεί με το θέμα της εκπαίδευσης, να ασκήσει εκπαιδευτική πολιτική στην Ένωση. Σήμερα η παιδεία, η εκπαίδευση είναι το κύριο είναι ε, ο κύριος κινητήρας για τη δημιουργία οικονομικής πολιτικής, πέρα από το να δημιουργούμε πολιτισμό κτλ. Ναι, έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ε, ποια μέτρα μπορούν να προετοιμαστούν για τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου, γιατί με την παλιά εκπαίδευση εμείς δεν κατορθώνουμε να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Ο κύριος Τάκουλα από την ε, Φινλανδία. δεν πρόκειται να κάνω ερώτηση. Ε, θα πέρασω στο διατάφτα. Δηλαδή, τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας για να βελτιώσετε την εκπαίδευση των δασκάλων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι, όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στην Ευρώπη να είναι σωστά εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να περνούν την παιδεία στα παιδιά. Θεωρείτε ότι κατά διάρκεια της ε, προεδρίας σας αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα. Πώς θα βελτιώσετε ακριβώς την εκπαίδευση των δασκάλων. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τις ε, εξηγήσεις που μας δώσετε για τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Εγώ συμφωνώ, όπως είναι και λογικό, νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικές και προτεραιότητες Προεδρίας αυτή στο θέμα της παιδείας. Ε, η παιδεία πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών και της οικονομίας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Εσείς ε, ήδη σχολιάσατε το πώς θα προσαρμοστεί η κατάρτιση ε, των ατόμων στις αναγκαιότητες της νέας αυτής οικονομίας που είπαμε ότι χρειαζόμαστε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Όταν μιλάμε για αυτή τη νέα οικονομία, για νέους οικονομικούς τομείς, μιλάμε πολύ για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ε, έτσι λοιπόν για το θέμα της ενίσχυσης δημιουργικότητας. Ε, το Κοινοβούλιο εκπώνησε πριν 1,5 χρόνο μία έκθεση για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών. Ε, αυτό αναφέρεται όχι μόνο, απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, αλλά ε, πρέπει να αποτελούν τα μαθήματα αυτά τμήμα των σχολικών προγραμμάτων ακριβώς ε, για να ενισχυθεί η δημιουργικότητα. Έτσι μιλάμε όταν για τις δεξιότητες, τις βασικές δεξιότητες ε, που θέλουμε να αναθεωρήσουμε ε, και αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε μεταξύ των προτεραιοτήτων και τη διδασκαλία αυτών των καλλιτεχνικών μαθημάτων προκειμένου λοιπόν να δώσουμε μία όθηση στη δημιουργικότητα. Bien, lo voy a intentar, Presidenta. Να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Θα προσπαθήσω. Οι καθηγητές έχουν τεθεί στο κέντρο του συστήματος ε, με την πεποίθηση ότι η πραγματική τροποποίηση του σημερινού καθεστώτος ε, της εκπαίδευσης ε, σήμερα περνά από την αναθεώρηση ε, και του καθεστώτος των ε, καθηγητών. Οι ερωτήσεις κατευθύνονται προς το τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη απέναντι στους καθηγητές, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάρτισή τους, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κινητικότητά τους. Ίσως ε, στο κέντρο αυτών των ερωτήσεων ε, υπάρχει και κάποιος στοχασμός, κάποιος προβληματισμός ότι μας μένουν πολλά ακόμα να γίνουν σε ένα χώρο που προσπάθησε με ορθά επιχειρήματα να πείσει τις εκπαιδευτικές κοινότητες. Ε, φαίνεται ότι πρέπει να προωθήσουμε τη συμμετοχή γιατί κάτι μάλλον δεν πηγαίνει καλά με το μοντέλο. Ε, ουσιαστικά πρέπει οι επιστημονικές κοινότητες να το αποδεκτούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε μηχανισμούς συμμετοχής αυτών των κοινοτήτων στη διαδικασία της Μπολόνια. Δεν θα υπάρχει ούτε Μπολόνια, ούτε νέος ευρωπαϊκός χώρος, αν οι καθηγητές και οι ε, εκπαιδευτικές κοινότητες δεν τα αποδεκτούν. Έτσι λοιπόν πρέπει να τους πείσουμε ε, και πρέπει να αναγνωριστεί η εμπλοκή τους ως κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα υπάρχουν ε, λιγότεροι δισταγμοί και φυσικά αυτό σημαίνει κάτι που έχουμε μάθει όλοι, ότι η Ευρώπη του πολιτισμού, της παιδείας, των πανεπιστημίων βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας. και μάλιστα αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο σε στιγμές οικονομικής κρίσης δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να ε, αναπτυχθεί η Ευρώπη γιατί δίχως κατάρτιση δεν υπάρχει απασχολησιμότητα, δίχως συγκεκριμένη κατάρτιση δεν υπάρχει μέλλον για την κινητικότητα. Εμείς θέλουμε να αναζητήσουμε στοιχεία κινητικότητας όμως οι αρμοδιότητες στην εκπαίδευση ε, οι στην εκπαίδευση δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρώπη. Είναι πιο πολύ πολύπλοκα τα πράγματα, όμως είναι βέβαιο ότι έτσι όπως δημιουργήθηκε εμπιστοσύνη στο θέμα της κινητικότητας των φοιτητών, αυτό πρέπει ε, να ε, συνεχιστεί και πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή που είναι η αυτονομία των πανεπιστημίων. Η αυτονομία των πανεπιστημίων είναι σημαντικό στοιχείο, καθαριστικό στοιχείο αυτής της κινητικότητας, γιατί ε, αν υπάρχουν υπάρχουν συμφωνίες. Αυτό επιτρέπει ένας καθηγητής να αναγνωρίζεται, να αναγνωρίζονται οι δεξιότητές του και οι ικανότητές του σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας. Όμως είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ ε, του να μην ε, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ σκέψεων που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ε, Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ βαθιά συνέργειες μεταξύ των δύο και αν ε, θέλουμε να αναφερθούμε στη στρατηγική για το 2020. Η ανταλλαγή απόψεων μας ε, βοηθά να προετοιμάσουμε την ε, νέα στρατηγική της Λισαβόνας. Έχουμε τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τυπική του Συμβούλια και προβλέπεται ότι θα υπάρχει έκτακτη συνεδρία στις 11 Φεβρουαρίου και στο Μάρτιο έτσι ώστε να ιδρυθούν τα περιφερειακά συμβούλια. όμω εμείς θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις στις συζητήσει αυτές και αυτό που μου φαίνεται ιδιαίτερα σαφέ είναι ότι αυτή η ιστορία της δημιουργία εμπιστοσύνη είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης. Και αν λέμε εδώ ότι θέλουμε να θέσουμε ε, τη γνώση στην καρδιά της νέας οικονομίας είναι γιατί έχουμε σχετική εμπειρία. Ε, είναι ότι ε, η οικονομία που δεν βασίζεται σε αξίες της εκπαίδευσης και του πολιτισμού δεν δημιουργεί ευημερία. δεν ε, θα υπάρχει καμία πραγματική διέξοδο από τη βαθιά κρίση αν στην καρδιά αυτής της κρίσης δεν θέσουμε τον πολιτισμό και την παιδεία ως καθοριστικούς παράγοντες ε, για την απασχολησιμότητα και την κατάρτιση. Ε, αναφερθήκατε και στη διδαχή των ε, καλλιτεχνικών ε, μαθημάτων. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να αποτελούν τα μαθήματα αυτά στοιχεία που προωθούν την προσωπική κουλτούρα και τη δημιουργικότητα. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να επιτρέψουμε να υπάρχουν καλλιτεχνικά μαθήματα, διδαχή καλλιτεχνικών μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Και φυσικά, ε, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης ε, των καθηγητών, θεωρώ ότι είναι καθοριστικά αυτά ε, στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης και εμείς Ε, ουσιαστικά δεν πρέπει εδώ να ε, λέμε ότι ε, οι καθηγητές έχουν μορφωθεί άπαξ και τέλος. θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο όπου θα υπάρχει κινητικότητα των καθηγητών και θα υπάρχουν και συγκεκριμένες δραστηριότητες κατάρτισης και θα υπάρχει και μόνιμη αξιολόγηση, διαβίω αξιολόγηση. Εγώ νομίζω ότι στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια πολλά πράγματα έχουν γίνει ορθά, όμως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αν δεν εμπλέξουμε ε, τους πρωταγωνιστές που είναι οι εκπαιδευτικές κοινότητες και οι καθηγητές, αν δεν δημιουργήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη που μόνο, γεννάται μόνο από την αυτονομία, ε, τότε πιθανότητα η διαδικασία της Μπολόνια δεν θα αποφέρει τους καρπούς που επιθυμούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις σας και αν ε, μετά υπάρχει χρόνος θα σας δώσω και πάλι το λόγο για να επανέλθετε εφόσον το επιθυμείτε. Κύριε Παλιαδέλη. Κύριε Επίτροπε, για... κύριε, Προ... Ε, κύριε Υπουργέ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε ό,τι αφορά ότι αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι η ομορφία στα πανεπιστήμια, αλλά η πολυμορφία η οποία όμως θα αντιμετωπίζεται με κριτήρια που θα επιτρέπουν την ε, ε, εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα ομολογουμένως, μια και είμαστε και Επιτροπή Πολιτισμού, να ακούσω λίγο παραπάνω για την άποψή σας για τις ανθρωπιστικές σπουδέ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πώς θα σκοπεύατε να τις υποστηρίξετε. Αλλά η ερώτηση που θα θέσω είναι ποια είναι η γνώμη σας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ειδικότερα ποια είναι η γνώμη σας για τον για το franchising των ιδιωτικών πανεπιστημίων, πώς δηλαδή αντιμετωπίζεται μια διαδικασία που είναι μια εμπορική, ε, εμπορική διαδικασία και πώς σκοπεύετε να τη μετατρέψετε, αν μπορείτε, ε, σε ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα διασφαλίσει την ποιότητα στη δημόσια ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Danke, Frau Trüppel, Frau Trüppel. Η Αντιπρόεδρος, κυρία Τρούπελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Η κυρία Πακ μετά την εισαγωγή της ε, είπε ότι φαντάζεται ότι θα μας στηρίξετε όταν ε, θα πρόκειται για την προαγωγή της ε, πολιτικής παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να την τοποθετήσουμε στο επίκεντρο της ε, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Δεν θέλω να γνωρίζω το εξής. Ε, εσείς θα κληθείτε να εργαστείτε με τη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού. Και τελικά τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι μπορείτε με αυτή τη στρατηγική να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των κρατών μελών. Και αν θελήσετε να διοχετεύσετε περισσότερα κονδύλια στην παιδεία, αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε την ανακατανομή στον προπολογισμό και αν το κάνετε αυτό, από πού θα κόψετε κονδύλια για να δώσετε στην παιδεία ή αν δεν σκοπεύετε να κάνετε αυτό, τότε πού θα βρείτε άλλα κονδύλια για να τα δώσετε. Επόμενος ερωτών. Κύριε Υπουργέ, από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, με το σύστημα της ε, παιδείας ε, αν δεν μπορούν οι ε, πολίτες ε, να βρουν θέση. Δεν ξέρω αν αυτό ε, σημαίνει ότι απέτυχε η διαδικασία της Μπολόνια ή μήπως απλά και μόνο είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην παιδεία και την πραγματική ζωή. Θα ήθελα λοιπόν ή δυνατόν να αναζητήσετε τους λόγους που διακοπή. Υπάρχει τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Δυστυχώς μας συγχωρείτε και εμάς υπάρχει κάποιο, κάποιο τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Δεν περνάει μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Λυπούμεθα πάρα πολύ. Πρόεδρος, δυστυχώς από ό,τι ακούστε υπάρχει ε, πρόβλημα αλλά σας καταλάβαμε στα ισπανικά. Από ό,τι φαίνεται μερικοί τα καταφέρνουν θαυμάσια με τα ισπανικά. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, να συνεχίσουμε. Λέει, πρόεδρος, λύθηκε το τεχνικής φύσεως πρόβλημα. Θα συνεχίσετε. Κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριο Μπίσκι, πρέπει να σας πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπατε σχετικά με τους ε, στόχους. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα που δεν γνωρίζω ε, πώς μπορεί κάτι να το λύσει και θα ήθελα να σας το επισημάνω. Αναφέρομαι στην ε, σχέση ανάμεσα στην παιδεία και την ένδυα. Η σχέση αυτή είναι όλο και πιο στενή. Η κοινωνιολογία της ε, παιδείας έχει εντοπίσει ότι η φτώχεια των παιδιών ορίζει και καθορίζει τη σταδιοδρομία τους, την επαγγελματική. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχέση ανάμεσα στην φτώχεια και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Αυτή η σχέση είναι πιο ισχυρή στη Γερμανία από άλλες χώρες. Υπάρχει όμως και αλλού. Κατόπιν τούτου υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα παιδείας, τα οποία όμως ε, θα μπορούσαν να αποτύχουν, γιατί ακριβώς ε, ορισμένα παιδιά δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το πρόβλημα, το φραγμό της φτώχειας. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Yes. Χωρίς μικρόφωνο, μάλιστα. Δεν ε, θέλουμε μια ομοιόμορφη Ευρώπη η ποικιλομορφία είναι συμβατή με τους κοινούς χώρες. Η διαδικασία της Μπολόνια δεν θέλει να εξαλείψει τις διαφορές των πανεπιστημίων των χωρών. Αυτό δεν είναι το ορθό μήνυμα. Το έχουμε κάτι κοινό σημαίνει ότι έχουμε συστήματα όχι μόνο συγκρίσιμα, ε, αλλά και συμβατά Η Ευρώπη είναι ένας ε, χώρος συνδύωσης ε, και υπάρχει κινητικότητα ακριβώ γιατί τα συστήματα έχουν παρόμοιες δομές και μπορούν να συγκριθούν. Όμως ε, αυτό κατά πολεμά έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι κάθε πανεπιστήμιο θα χάσει την ιδιαιτερότητά του. Το αντίθετο λέμε ότι κάθε πανεπιστήμιο θα έχει τις δικές του στρατηγικές, τα δικά του ίδια χαρακτηριστικά Απλώς ε, θέλουμε εδώ να δημιουργήσουμε ένα χώρο ανταγωνιστικότητας και ξεχρονισμού. Ε, τώρα για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές θα ήθελα να πω ότι η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη και το λέω γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Φαίνεται ότι η οικονομία είναι μόνο μία τεχνοκρατικού χαρακτήρα επιστήμη όμως έχουμε και την ανθρώπινη διάσταση της γνώσης, τη διάσταση του πολιτισμού σε σχέση με τη γνώση, κάτι καθοριστικό. Όμως ε, σε ένα μοντέλο υπερβολικά τεχνοκρατικό ξεχνάμε πολλές φορές ακριβώς ε, το πόσο ε, συνεισφέρει η ανθρωπιστική, η ανθρώπινη πτυχή ε, και έχουμε την λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και άλλες επιστήμες που πραγματικά αποτελούν την καρδιά της πραγματικής ταυτότητας της Ευρώπης και δεν είναι ορθό το μήνυμα, ε, να θεωρούμε τις ανθρωπιστικές σπουδέ ως σπουδέ που δεν έχουν ε, αποδοτικότητα, γιατί πρέπει να μιλάμε για κοινωνική αποδοτικότητα, για κοινωνική κερδοφορία. Και αυτή είναι τεράστια και αυτό δεν συγκρίνεται με την οικονομική κερδοφορία. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό ή στην κλίμακα των αξιών μας να ξέρουμε ότι η κοινωνική κερδοφορία και η οικονομική κερδοφορία είναι συμβατές και επομένως ε, πρέπει να πούμε ότι δεν ε, πρέπει να γνωρούμε ε, τα αιτήματα της κοινωνίας και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί σε κάποια από τις ερωτήσεις που έγινε. Δηλαδή, ρωτήθηκε γιατί δεν ε, υπάρχουν κάποιες ε, απαντήσεις, δεν υπάρχει ανταπόκριση, παραδείγματο χάρη, ε, όταν υπάρχει αίτημα για συγκεκριμένες σπουδές. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε να προωθήσουμε αυτές τις σπουδές. Επίσης, όταν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρτιση και παιδεία, έχουμε μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Όσοι έχουν καλύτερη κατάρτιση παραμένουν περισσότερο στο χώρο εργασίας και αν χάσουν την εργασία τους, τότε είναι πιο εύκολο να ξαναβρούν δουλειά. Γιατί δεν θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι η αποσχολησιμότητα δεν έχει να κάνει με την κατάρτιση. Το αντίθετο, ξέρουμε ότι όταν έχουμε καλύτερη και πιο ποιοτική κατάρτιση υπάρχει και μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Όμω ε, έγινε μία μελέτη για του ε, τεχνικού λόγου που οδήγησαν ε, ορισμένα πτυχία, ορισμένες σπουδές δεν βρίσκουν στη συνέχεια διέξοδο στην αγορά εργασίας θα ήταν ενδιαφέρον από τη σκοπιά της αυτονομίας των πνευστημίων αυτές οι σπουδές να ανταποκρίνονται, οι νέες σπουδές, τα νέα πτυχία να ανταποκρίνονται στα κοινωνικά αιτήματα. Τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν ε, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί τρόποι να οργανωθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ε, δεν ε, θεωρώ ότι ούτε εδώ πρέπει να μιλάμε για μια ομοιόμορφη εικόνα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν διαφορετικέ νοοτροπίε ε, και οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι επικεντρώνονται περισσότερο στην οικονομία, ενώ άλλα πανεπιστήμια έχουν διαφορετική νοοτροπία. Ε, Όμω πρέπει να εγγυθούμε διότι να μοντέλα ε, χρηματοδότηση του συστήματο των πανεπιστημίων που να επιτρέπει μεικτές ε, φόρμουλες χρηματοδότησης και αυτές οι μεικτέ μορφές πρέπει να υποστηρίζουν κάτι που θεωρούμε θεμελιώδες το ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και ως δημόσιο αγαθό πρέπει να το εγγυώνται τα κράτη, πρέπει να είναι δικαίωμα των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν συστήματα συμβατά που μπορούν να συμβιώνουν και με άλλε μορφέ πανεπιστημίων. Όμω τι είναι ένα πανεπιστήμιο. Αυτό είναι θεμελιώδες ερώτημα στην Ευρώπη. Τι χαρακτηρίζει ένα πανεπιστήμιο. Ε, ποιες ε, απαιτήσει πρέπει να πληρούνται. Ε, τι δημόσιο λειτουργήμα, ποια δημόσια λειτουργία πρέπει να πληρεί ένα πανεπιστήμιο και ποιε ποιοτικέ εγγύσει πρέπει να παρέχονται σε ό,τι αφορά του καθηγητές και τις ποιε χρηματοδότηση. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα θέματα. Ε, Δηλαδή, μεταξύ των πρεπιστημίων που είναι ποιοτικά και επιτελούν δημόσιο έργο και μεταξύ αυτών που δεν το πράττουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά με ε, το θέμα της ε, χρηματοδότησης, ε, εγώ θεωρώ ότι η χρηματοδότηση και η παιδεία αποτελούν ε, σημαντικό κεντρικό άξονα ε, στη στρατηγική. Εμείς θα βρούμε μια λύση για τη χρηματοδότηση και επίσης μπορούμε να ανοίξουμε και τη συζήτηση για νέους πόρους. Αλλά αν η παιδεία δεν τεθεί στο κέντρο της στρατηγικής, όχι μόνο έχουμε θεωρητικό πρόβλημα, αλλά έχουμε και πρόβλημα χρηματοδότησης. Και επομένω, ο στόχος μας καταρχήν είναι να πετύχουμε αυτή την παρέμβαση, αυτή την παρουσία αν θέλετε, εγώ ε, αναφέρθηκα στο θέμα της ανέχειας και είπαμε ότι η παιδεία είναι η πρώτη κοινωνική πολιτική και ε, ουσιαστικά ε, η παιδεία ε, συνεισφέρει τα μάλα για την κοινωνική ένταξη. Η ισότητα των ευκαιριών, ε, η παιδεία, η ανώτερη εκπαίδευση συνεισφέρουν στην ε, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Και εγώ πιστεύω ότι οι λόγοι είναι και κοινωνικοί, όχι μόνο εκπαιδευτικοί και σε ό,τι αφορά την αποτυχία. Και μιλάμε ε, για ανέχεια που δεν είναι μόνο οικονομική. Εγώ νομίζω ότι για να βγει κανείς από τη φτώχεια, ο καλύτερος δρόμος είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Αυτό στην έκθεση του ΩΣΑ ε, ορίζοντας του 2020 και λέγεται ότι μέσω της παιδείας μπορεί να αποτελεσματικά αυτή η ανέχεια, αυτή η φτώχεια. Yes. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε ε, Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένας με όσα μας είπατε. Αυτό όμως που ίσως δεν είπατε είναι κάτι που σχετίζεται με την έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των πανεπιστημίων Αφενό και των επιχειρήσεων αφετέρου στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη στρατηγική αυτή που ε, προτείνεται, πιστεύουμε ότι η παιδεία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται να αποφύγουμε να υπάρχει ένα πολιτιστικό όριο μεταξύ της ε, των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων, όπως ελεγχθεί ήδη. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να κάνουμε κάτι περισσότερο μέσα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σκουρία. Ε, Ευχαριστώ. Πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι μου άρεσε που αναφερθήκατε στην προτεραιότητα που θέλετε να δώσετε στην παιδεία η Ευρώπη της γνώσης ε, είναι ε, ως όρος πάρα πολύ κατάλληλος και στοχευμένος και επίσης ε, μπορούμε να αναφερθούμε και ε, στο ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα που θέλετε να δώσετε στη δράση σας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, ήταν ήδη ξεκάθαρα τα μέσα προσιοθέτηση για το περιορισμό ή εξάλληψη ενός φαινομένου που εμφανίζεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη και αφορά το διασκορπισμό και την εγκατάλειψη των σχολείων. Και δεύτερον, θα ήθελα να φερθώ και σε ένα θέμα που συζητήθηκε και από άλλες επιτροπές και έχει να κάνει ε, με την πραγματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα, ένα άνθρωπο, ένα άτομο που σπουδάζει νομική στην Ισπανία, έχει δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμά του, ε, παραδείγματο χάρη νωρίτερα σε σχέση με έναν Ιταλό ε, υπάρχουν πραγματικά συγκεκριμένα εμπόδια ε, για να μπει κάποιος στο χώρο εργασίας σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ενώ αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, έχει σπουδάσει στην Ισπανία, ε, νομική δυσκολεύεται λιγότερο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου απαντήσετε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, Ιβάν. Σας ευχαριστώ. Απαντήσετε στις μισές από τις ερωτήσεις μου, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να επαναλάβω όμως μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει κάποιο πολύ συντηρητικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δεν προσαρμόζονται δηλαδή στις ανάγκες της οικονομίας εύκολα. Δεν θα σας ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο προβλέπετε εσείς η υιοθέτηση μέτρων που θα μπορούσαν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα να καθιστούν πιο ευέλικτα, ιδίως τώρα που έχουμε μια οικονομική και κλιματοπιστική κρίση και η αγορά εργασίας αναδιοργανώνεται συνεχώς και υπάρχουν πολλοί εκπαιδευμένοι από πανεπιστήμια ή και κατατισμένοι σε κάποια εργασία που δεν θα μπορούν να βρουν μια δουλειά στον τομέα για τον οποίο έχουν εκπαιδευτεί. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν ανησυχείτε από την άλλη μεριά που υπάρχουν τόσες επιχειρή... ε, κυβερνήσεις που προσπαθούν να περικόψουν τα κονδύλια για την παιδεία για να μειώσουν το δημόσιο έξοδο. Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εξαιρετικοί κύριοι βουλευτές. Πράγματι, το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να είναι ένας χώρος διδασκαλίας και διαβίβασης της γλώσσης, αλλά πρέπει να είναι και ένας χώρος δημιουργίας της γνώσης και έρευνας. Τα τελευταία δέκα χρόνια μάθαμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει και ένα τρίτο καθοριστικό λειτουργήμα του Πανεπιστημίου μέσα στο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή η διαβίβαση της γνώσης στην κοινωνία και πρέπει να επιστρέφουμε την γνώση στην κοινωνία, δημιουργώντας έτσι ευημερία για τις ε, χώρες. Το Πανεπιστήμιο δεν ε, ε, πρέπει να περιορίζεται, αλλά πρέπει να διαβιβάζει και τη γνώση αυτή και αυτό σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο συνδέεται πάρα πολύ με το τι υπάρχει γύρω του σε κοινωνικό, επιχειρηματικό, περιφερειακό επίπεδο. Ένα πανεπιστήμιο πρέπει ουσιαστικά ε, να εμπλέκεται ε, στο ευρύτερο πλαίσιο αν το Πανεπιστήμιο εμπλέκεται θα πρέπει να σχεδιάζει όλες τις δραστηριότητες στα πλαίσια αυτά και θα πρέπει και το ίδιο να έχει επιρρηματικό πνεύμα, θα πρέπει να έχει αυτή την επιχειρηματική νοοτροπία. Όχι μόνο να συναντάτε με τους επιχειρηματίες και τελευταία ε, ουσιαστικά είδαμε και μία αμοιβέληψη εμπιστοσύνη μεταξύ Πανεπιστημίου και επιχειρηματικού κόσμου. Ε, γιατί ο επιχειρηματικό κόσμο θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο ήταν πολύ επικεντρωμένο στον εαυτό του ε, και πολλοί ε, από το χώρο των πανεπιστημίων ε, κοιτούσαν με καχυποψία τον επιχειρηματικό κόσμο και θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κοινωνικό ενδιαφέρον από την πλευρά του σήμερα. Θέλουμε εμεί να προτείνουμε κοινού στόχου και να υπάρχει συνεργασία Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι ο επιχειρηματικό κόσμος ε, ουσιαστικά απλώ ε, παράγει κέρδο, ε, αλλά αποτελεί και ένα κόσμο πλούτου. Θεωρώ ότι πρέπει να προσδώσουμε κίνητρα στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να λειτουργήσουν ω διαβιβαστές τη γνώσης. Αν θέλουμε να είμαστε σε μια κοινωνία της γνώσης, πρέπει να δεικτούμε ότι η γνώση είναι η μεγαλύτερη αξία οικονομική και πολιτική και αν θέλουμε η ε, μεγαλύτερη κοινωνική δράση να συνδέεται ε, με τη γνώση, τότε θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία. Ε, θέλουμε τη γνώση αυτή να την καταστήσουμε καθολική Θέλουμε να διασκορπιστεί η γνώση που έχει επιτευχθεί ε, ήδη στις ε, οικογένειες, στα πανεπιστήμια όμως υπάρχουν, υπάρχει και τίμημα σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και διαδικασίες ποιότητας, ε, διαδικασίες αριστείας. Κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία ε, έχουν ε, ουσιαστικά ε, δημιουργήσει κάποιους διαγωνισμούς και εμείς πρέπει να εγγυθούμε να υπάρχουν υποτροφίες, να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στους τόπους αυτούς μάθησης. Αναφερθήκατε στο δίκαιο. Υπάρχουν πάρα πολλά ληφητητές ε, νομικοί στην Ευρώπη. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε ποια είναι τα κοινωνικά αιτήματα και σε σχέση με αυτά τα κοινωνικά αιτήματα ε, να ε, κάνουμε κάποια συγκέντρωση, αν θέλετε, πανεπιστημίων, στόχων κτλ. Όχι συγχώνευση πανεπιστημίων. Δεν αναφέρομαι στην συγχώνευση των πανεπιστημίων και το θέμα τη ισοδυναμία είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόβλημα. Και αυτό τόσο πολύπλοκο χαρακτήρα ε, έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά δικαιώματα, όχι μόνο με ακαδημαϊκά θέματα, γιατί πέρα από τα ακαδημαϊκά θέματα έχουμε και τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν και εκεί πρέπει να πετύχουμε την ομοιομορφία, την ομοιογένεια. Εγώ δεν νομίζω ότι τα συστήματα μας πρέπει να είναι πιο ευέλικτα μάλλον πρέπει συγγνώμη τα συστήματα μας να είναι πιο ευέλικτα, γιατί τώρα είναι ιδιαίτερα άκαμπτα. Ε, επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προσαρμοστικότητα των πανεπιστημίων. Σήμερα δεν βγαίνει κάποιο ε, από το Πανεπιστήμιο και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τι ε, προκλήσει. Ε, πρέπει να έχει τι ικανότητες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να μπορεί να προσαρμοστεί στι απαιτήσει και κάθε φορά θα πρέπει να προσαρμόζει τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. κάποτε θεωρούταν ότι η κατάρτιση που λαμβάνει κάποιον ίσχυε για όλη του τη ζωή. Ε, και δυστυχώς αυτό μας οδήγησε σε πολύ μεγάλη έλλειψη απασχολησιμότητας. Να σας πω ότι εμείς προτείνουμε επίσης την αναγκαιότητα να υπάρχει μεταρρύθμιση των ε, προγραμμάτων, να υπάρχει ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης από τα πανεπιστήμια και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή μοντέλου, ενολογική αλλαγή που θα θέσει την παιδεία στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Αυτό, αν το πετύχουμε σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Αβώνας και αν έχουμε τα ορθά επιχειρήματα, τότε είμαι σίγουρος ε, ότι ε, θα καταφέρουμε να βρούμε τη λύση στην εξίσωση και θα βρούμε και την ορθή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Δύο συνάδελφοι έχουν ακόμα ζητήσει το λόγο και δύο συμπληρωμικέ ερωτήσει υπάρχουν. Καταρχήν, κυρία Ανιμπάλ. Τα κυρία Χίρ και μετά οι δύο συμπληρωμικέ ερωτήσει, Τάκουλα και Μπαλιαντέλη. Καταρχήν κύριε Χάνιμπαλ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Σα καλωσορίζω κύριε Υπουργέ. Συζητάμε για την Πολόνια και την επαγγελματική κατάρτιση και την κινητικότητα των φοιτητών αλλά και των διδασκόντων. Εγώ θα ήθελα να θέσω το θέμα της ε, ε, εκμάθησης των γλωσσών στα σχολεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κινητικότητα, γιατί οι φοιτητέ και οι διδάσκαλοι τους δεν θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα εάν δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν ε, πληρεί το πρότυπο των δύο συμπληρωματικών ξένων γλωσσών. Υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως ξέρω, και θυμάμαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ε, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα δικά σχόλια, πώς θα το πετύχετε αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Χίρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τονίσατε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και ότι εδώ θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Το χαιρετίζω αυτό εγκαρδιότατα. Είπατε και ο ίδιος ότι είναι σημαντική η κινητικότητα και βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχουν πολλές ε, οικογένειες με κινητικότητα και ότι οι οικογένειες λόγω της κατάστασης ε, της απασχόλησης ζουν μερικά χρόνια στην Ιταλία, μερικά στην Αγγλία, μερικά στη Γαλλία. Τα παιδιά όμως πρέπει να πάνε και στα σχετικά σχολεία. Και θέλω να αναφερθείτε λοιπόν λιγάκι και στην κινητικότητα για τους μαθητές. Τα παιδιά δηλαδή αυτά των εργαζομένων, όταν ε, οι γονείς τους πάνε από τη μία χώρα στην άλλη, θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των σχολείων. Ε, θα ήθελα να ξέρω, σκοπεύετε εσείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να εκινήσετε μια πρωτοβουλία για να προωθήσετε αυτή την ιδέα του ενιαίου σχολείου Δηλαδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα σχέδιο με ένα πλαίσιο, με συνδυασμούς ε, των διαφόρων ε, μαθημάτων, ούτω ώστε ένα παιδί που ξεκινάει σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό, θα ήθελα το πω σχολείο, να μπορεί να συνεχίσει σε μια άλλη χώρα. Θα είχαμε επικουρικότητα γιατί τα κρατικό μέλη θα ακολουθούσαν κάτι τέτοιο εθελοντικά, από την άλλη μεριά όμως θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη αυτά τα ενδεικτικά, αν θέλετε, τα διπλώματα που θα είχαν τα παιδιά από το ένα σχολείο να αναγνωριστούν στο άλλο. Δηλαδή να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ιδέα, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ευρωπαϊκού σχολείου για να μπορούν να γνωρίζονται τα εκάστοτε διπλώματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπενεράτου έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προοπτικές που μας ανοίξατε. Τονίζοντα και θέτοντα στο επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική το θέμα τη παιδεία, Σημείωσα με ενδιαφέρον τη σημασία που αποδίδεται στα ανθρωπιστικά, στο ανθρωπιστικό κλάδο. Γιατί είπατε ότι αυτό είναι κάτι που εκπαιδεύει τον πολίτη ως πολίτη αναφερόμενο στην παιδεία όμω και στην νεολαία, δεν αναφερθήκατε καθόλου στην ενσωμάτωση των πιο ηλικιωμένων γενεών. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις στην ε, πολιτική των ανθρωπίνων πόρων αντιμετωπίζουν μια έναν ανταγωνισμό, αν θέλετε, μεταξύ της πρόληψης πρόσληψης συγγνώμη, νέων και πρόσληψης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Πώς θα βγει κανένα από το δίλημα αυτό και να υπάρχει μια πολιτική διαφορετική όσον αφορά την παιδεία και την κατάρτιση. Πώς αυτό που σήμερα είναι ένα πρόβλημα θα αποτελέσει πλεονέκτημα της πολιτικής για το μέλλον. Θα σας ευχαριστώ. Σύντομα, ο Άννα Τάκουλα, πολύ σύντομα μίλησες ήδη. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να επισέλθω εις βάθος στο θέμα που έθιξα προηγουμένως για την εκπαίδευση των διδασκόντων. Ξέρετε, Υπουργέ, ότι τα αποτελέσματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την βασική εκπαίδευση των παιδιών κατέδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ στα διάφορα κράτη-μέλη. Δείτε, παραδείγματο χάρη, τα αποτελέσματα των μελετών PISA Βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και στον τομέα της εκπαίδευσης των διδασκάλων όταν μιλάμε για την βασική εκπαίδευση των παιδιών. Βέβαια, την κυρία ευθύνη εδώ έχουν τα κράτη-μέλη. Αλλά εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι και στο ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι θα πρέπει να γίνει. Πιστεύει η Ισπανική Προεδρία ότι πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι για την εκπαίδευση των δασκόλων. Πώ θα το θέσουμε αυτό, παραδείγματο χάρη, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματο για το 2020. πώ θα βελτιώσουμε εκεί την εκπαίδευση των διδασκάλων που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των παιδιών μα για να έχουν όλε τι ίδιε ευκαιρίε. Ευχαριστώ, σύντομη κυρία Παγιαντέλη και μετά ο υπουργό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ίσως δεν έγινε απολύτω σαφή η ερώτησή μου που αφορά στη δημιουργία παραρτημάτων πανεπιστημίων, κύριε Υπουργέ, ε, από πανεπιστήμια σε άλλε χώρε. Το franchising. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τα franchising ε, γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. It's your turn. Η σειρά σα. Ευχαριστώ πολύ. Yo, yo creo que... Ναι, νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα σε σχέση με τις γλώσσες ε, και σε ορισμένες χώρες ε, παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό και στην Ισπανία υπάρχουν ε, προβλήματα. Βέβαια υπήρξε σημαντική βελτίωση, όμως πολλές φορές μιλάμε για γλώσσες ε, που μιλούνται από πολλούς ε, ανθρώπους και ε, αυτό μπορεί να μας έχει επιτρέψει αφενός να θεωρούμε ότι είμαστε καλυτερτές αλλά από την άλλη μας έχει περιορίσει στην κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θεωρούμε ότι η στρατηγική 2020 ε, πρέπει να θέτει όχι μόνο το θέμα της μάθησης των γλωσσών, αλλά και της διαβίου μάθησης και της πρόθεσης της ε, ισότητας ε, των ίσων Μιλήσαμε για όλα αυτά, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε καθοριστική προτεραιότητα. Μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσει ε, γίνεται λόγο ε, και για δίγλωσσα σχολεία. Ε, νομίζω ότι κάποιο το να γνωρίζει πάρα πολύ καλά μια γλώσσα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ανοίγονται και νέε δυνατότητε. Όμω, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασική η γνώση των γλωσσών και επίση ε, θεωρώ, και αυτό φάνηκε και με το πρόγραμμα Erasmus, ότι ε, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη γνώση της γλώσσα όταν κάποιο μεταβαίνει σε μια άλλη χώρα. Όμω ε, και η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί σε άλλε χώρε διαφέρει η κατάσταση, γιατί από την πρώτη στιγμή έχει προωθηθεί η διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η έννοια της κινητικότητας ε, είναι μία από τις πιο καθοριστικές έννοιες, αλλά όχι μόνο από τη σχολική σκοπιά, αλλά και από την κοινωνική και έχει να κάνει με την αποδοχή του άλλου ε, και θεωρώ ότι το Εράσμους έχει κάνει πολύ περισσότερα για την Ευρώπη από πολλούς ε, λόγους. Αυτό συνεισφέρει και ε, στην αναγνώριση, στη γνώση των άλλων. Δηλαδή είχαμε 4 εκατομμύρια ε, φοιτητών ε, οι οποίοι μετέβησαν σε άλλες πόλεις, γνώρισαν άλλους τόπους και άλλους ανθρώπους. Αυτή η κινητικότητα λοιπόν αποτελεί πολύ μεγάλη αξία και υπερβαίνει την ε, σχολική πτυχή. Η έννοια του Ευρωπαϊκού Σχολείου θεωρώ ότι τώρα δεν θα ανταποκρινόταν ε, στο ε, μοντέλο της ποικιλομορφίας και της συμβατότητας των συστημάτων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε συμβατά συστήματα, όχι ε, ταυτόσιμα συστήματα, ομογενή συστήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κάνουμε τα πράγματα ορθά. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι οι τρόποι αυτοί να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Το να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την παιδεία με την κατάρτιση είναι ζωτικό ε, η ένταξη των πιο ηλικιωμένων είναι επίσης ε, πολύ σημαντική. Εμείς ε, αναμένουμε η πρώτη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης 2014-2020. Θα συμπεριλάβει και θέματα που αφορούν τη διαβίου μάθηση. Και αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι διαρθρωμένα, δηλαδή ένα άτομο, μάλλον όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να προσφέρουν τόσο προγράμματα κατάρτισης και διαβίου μάθησης. Και ελπίζω αυτά τα προγράμματα της διαβίου μάθησης να μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Τώρα για τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ δεν θέλω να ανοίξω μια νέα συζήτηση, καθώς ε, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, κάποια στιγμή, ε, πέρα από το να συγκρίνουμε τα μοντέλα, να δούμε ποιες είναι και, ποια είναι και τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε. Η έννοια της εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας, δεν είναι ταυτόσιμη σε όλες τις χώρες. Πολλές φορές συγκρίνουμε αυτά τα μοντέλα, ενώ ξεκινάμε από διαφορετικές έννοιες. Όμως ε, εγώ ήθελα να πω ότι πρέπει ε, να είναι ζωτικής σημασία η κατάρτιση των καθηγητών και Πρώτη φορά ε, απαιτήθηκε φέτος ε, στην Ισπανία για τους καθηγητές να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού θα μπορούσαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο επιτυχιακό για την κατάρτιση των καθηγητών. Γιατί ε, υπάρχει πεποίθηση ότι η κατάρτιση των καθηγητών και το σύστημα ε, της ε, επιλογής των καθηγητών πρέπει να την χάνουν συγκεκριμένου ελέγχου. Εμείς ε, ως ε, χώρα αυτή τη στιγμή έχουμε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά Θέλουμε να σκεφτούμε με σοβαρότητα ποιο θα είναι το βεληνικές που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο όραμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το franchising, ε, εγώ μπορώ να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι δεν αγοράζεται ούτε πολύ η παιδεία και επομένως ε, πρέπει να <laughs> βρίσκεται στο περιθώριο μιας ε, αγοράς αγροπολισίας, αν θέλετε. Και εγώ πιστεύω σε ένα ανοιχτό ε, χώρο με ε, πολλαπλές φωνές. Εγώ δεν πιστεύω ότι η παιδεία και η εκπαίδευση είναι εμπόρευμα, ούτε πιστεύω ότι η εκπαίδευση ως τέτοια πρέπει ε, να περιγράφεται με όρους όπως πελάτης, προϊόν, κατανάλωση. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης και επομένως ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε και κάποιους κανόνες ρύθμισης ε, έτσι ώστε να είναι ε, συμβατή η ελευθερία της κινητικότητας αλλά να μην μπούμε και σε μια λογική αγοροπολισίας πτυχίων. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και η Ευρώπη πάντοτε πίστευε ότι ο πολιτισμός και η παιδεία ουσιαστικά προωθούν την προσωπική αξιοπρέπεια και την κοινωνική αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι μας απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις. Σχεδόν ακρόαση ήταν αυτό που κάναμε μαζί σας. αλλά βρήκαμε μαζί σας νομίζω ένα συμπολεμιστή, αν μπορώ να το πω έτσι, και ελπίζω και με την, γενικά με την Ισπανική Προεδρία. Και άμα λέτε ότι περισσότερα πέτυχε το Erasmus από πολλά περισσότερα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι το πρόγραμμα Κομένιους διδρύθηκε επειδή ακριβώς ήταν τόσο επιτυχές το πρόγραμμα Erasmus και το Γκρούντ είχε επίσης για τον ίδιο λόγο για την ε, εκπαίδευση των ε, ενηλίκων. Και ελπίζω θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε όλα αυτά τα προγράμματα και το Λεωνάρντο βέβαια που έχει ένα δικό του στυλ. Τούτων εχθέντων, δεν θα προσθέσω και κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Είπατε ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι πιο ευρωπαϊκά. Εγώ έχω να πω ότι ήδη το Μεσαίωνα ήταν ευρωπαϊκά τα πανεπιστήμια. Εμείς τα καταντήσαμε εθνικά. Εμείς τα εθνικά κράτη τα περιορίσαμε, δημιουργήσαμε εμπόδια και γι' αυτό θα ήμουν πολύ ευγνώμη με τη βοήθεια της Μπολόνια εξαλείψουμε τα εμπόδια αυτά που υπήρχαν. Και στην επόμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη νομίζω για το θέμα της Μπολόνια να φροντίστε μαζί με τους συναδέλφους τους να ασχοληθείτε ακριβώς με την εξάλληψη αυτών των εμποδίων. Γιατί σας λέω, τα πανεπιστήμια στο παρελθόν ήταν ευρωπαϊκά, αλλά από πολλούς υπαλλήλου και υπουργεία ε, μετατράπηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις ιδέες κάθε κράτος. Και η Μπολόνια αν έχει ένα στόχο θα πρέπει ακριβώς να κατακτήσει πάλι δυνατή την κινητικότητα που ήταν δυνατή το μεσαίωνα. Λοιπόν, θα ήταν καλό έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με στα πλαίσια της Μπολόνια. Θα ήμασταν ευγνώμενες γι' αυτό και θα δούμε στο τέλος της Προεδρίας σας πόσο προχωρήσαμε από κοινό. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, καλή τύχη και σας διαβεβαιώ ότι εκεί που χρειαζόσατε τη βοήθειά μας θα σας προσφέρουμε ευχαρίστως. Και θα ήθελα να σας πω ότι οι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται και πάρα πολύ να προσκληθούν σε οτιδήποτε οργανώ... εκδήλωση οργανώσετε στο παρελθόν πολλές προεδρίες ξεχνάνε ότι υπάρχουν και οι ευρωβουλευτές που τις χρειαζόστε για τη συναπόφαση. Ελπίζω να είναι μια θαυμάσια εξαίρεση η Ισπανία. Σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ συναδέλφους. Θα αποχαιρετήσουμε τον Υπουργό. Θα διακόψουμε πολύ σύντομα τη συνεδρίαση. Υπάρχει και ένα τεχνικό πρόβλημα και θα πρέπει να διορθωθεί.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 We start once again. The technical problems are solved, I was told. Λοιπόν, μου λένε ότι λύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα. Σας παρακαλώ. The people of the administration of the sick. Παρακαλώ, να σταματήσετε συνομιλίες. Θα θέλουμε να εργαστούμε εδώ. Καθίστε στις θέσεις σας κύριε Μπερλιγκέρ, με που ήρθατε. half of Spain was here. Okay. <laughs> So, es geht weiter in Deutsch. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Σημείο 5 σήμερα τη διάταξη. Κατάσταση μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ψηφιακή τεχνολογία από το E2010 στο Digital EU. Η συζητήση μα είναι ο κύριο Ιβάν. Θέλω να παρουσιάσει βέβαια την γνωμοδότησή του επί επιτροπή έχει αλλάξει το τίτλο. Η κυρία Δεκαστήλιο μετενόμασε την έκθεση αυτή που λέει ορίζεται μια νέα ε, ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη από το E2010 στο Digital EU. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια και τίποτα. Θα ακούσουμε την, την δική σας γνωμοδότηση, αγαπητέ Ιβάν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η γνωμοδότηση αφορά εκείνες τις πτυχές για τις οποίες είναι αρμόδια η δική μας επιτροπή. Δεν είναι δηλαδή μια συνολική προσέγγιση. Εκτός αυτού είναι μια εργασία αυτή τη στιγμή που συνεχίζεται και γι' αυτό θα χαρώ πολύ για τις συμβολές των συναδέλφων. Για όλους μας και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες η επιτάχυνση της ε, ε τεχνολογίας στον ε, το, τομέα αυτό είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Ζούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε καθημερινά με τη βοήθεια των ψηφών αυτών των τεχνολογιών. Όμως η στρατηγικη η E2010 δεν μπόρεσε να οδηγήσει στα αποτελέσματα που θέλουμε. Άλλοι στόχοι έχουν επιτευχθεί βέβαια, άλλοι καθόλου. Θα ήθελα στους επιτευχμένους να πω ότι η ανάγκη της βελτίωσης της ε, ποιότητας ζωής και της αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν κατάφερε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα. Προφανώς χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική. Και είναι προφανές ότι η νέα αυτή στρατηγική θα πρέπει στα σημεία κίνησης να έχει εκείνους τους στόχους που δεν έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής με τη στρατηγική ή 2010. Η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευρεία και θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνοι θα πρέπει να ωφεληθούν κυρίως από την πολιτική μας. Μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Θα πρέπει να τονίσουμε την ποιότητα της πληροφορίας, την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις πτυχές που αφορούν την ασφάλεια της ε, πληροφόρησης. Επίσης, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να βοηθήσουν την Ένωση να γίνει πιο αναγωνιστική σε διεθνό επίπεδο και να πετύχει μια οικονομία βασιζόμενη στις γνώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τεχνολογίες αυτές να υποστηριχθούν οι ανάγκες των πολιτών. Η γνωμοδότησή μου συμπεριλαμβάνει τρία σημεία που κατά γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, είναι ουσιαστικό να αναπτυχθεί η δυνατότητα της νεολαίας να χρησιμοποιεί τους ε, δυνατότητες της πληροφορικής. Και έχουμε εδώ το e-learning και το e-government. Οι τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν τις ικανότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά απασχόλησης ή στην προσαρμογή της πραγματικότητας της κοινωνίας καθημερινά. Επίσης, με το e-government θα μπορούν οι νέοι γλίγορα να έχουν τη δυνατότητα να χειριστούν αυτές τις δυνατότητες που τους η τεχνολογία. Και αυτά τα μέτρα υποστηρίζουν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου βασιζόμενη στις γνώσεις. Θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία της προσέγγισης αυτής, της ε, ε, προσέγγισης Ευρωπαϊκής και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι συμπληρωματική του Google. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός με τα Google Books γνωρίζω τις νομικές δυσκολίες που θα έχει αυτή η κατάσταση και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πύλη που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες δηλαδή, βιβλία, και ξεκινώ από την ε, δήλωση του Ζωμονέ ότι αν ξαναμελετήσουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πολιτισμός σαν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των κρατών. Πιστεύω ότι ε, η πολιτιστική πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής αυτότητας και μια τέτοια πύλη θα μπορούσε να επιτρέψει την επίτευξη της δυνατότητας ε, κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό άσχετα που ζει. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αισθανόμαστε κάθε μέρα ότι είμαστε Ευρωπαίοι και πολίτες της Ευρώπης. Τέλος πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τις προηγμένες υπηρεσίες ε, ICT θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να μάθουν περισσότερο όσον αφορά τα ωφέλη των τεχνολογιών αυτών και ταυτόχρονα θα τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς θα μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές. Και εδώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μία δυνατότητα ανάπτυξη μιας εκστρατείας που θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβαση. Παραδείγματος να έχουμε ένα ετήσιο βραβείο για το καλύτερο ετήσιο σχέδιο. Εδώ θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο νομίζω. Αυτές είναι λίγες πτυχέ που θα ήθελα να σας παρουσιάσω όσον αφορά αυτή την ε, γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι η στόχοι της στρατηγικής ή 2010 ήταν καλή. Τα επιτεύγματα μέχρι στιγμή είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξου στόχου για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Τρούπελ, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφε Ήβαν, από αυτά που μας είπατε, εγώ κατάλαβα ότι οι στόχοι σας είναι ιδιαίτερα ευρωπαϊκή, με την έννοια ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να συμπεριλάβετε τους πολίτες, κυρίως ε, τους ε, νέους ε, και να τους προσφέρετε τις δυνατότητες μέσα από την πληροφορική. Θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις για θέματα που δεν τα κατάλαβα καλά, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μπίσκι, γνωρίζουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Γερμανία, υπάρχει το πρόβλημα της παιδείας και της φτώχειας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εσείς τώρα είπατε ότι επιθυμείτε την ε, τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας να την ε, προσφέρετε κυρίως ε, στα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ έχω κάνει εμπειρία ότι τα παιδιά αυτά τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από τους γονείς τους, πόσο μάλλον από τους ηλικιωμένους. Άρα δηλαδή θέλουν να εξοικειωθούν με κάποια θέματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Βεβαίως το να τους προσφέρει κανείς την τελευταία τεχνολογία, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και από ό,τι έχω κάνει κάνει την εμπειρία, δεν ξέρω αν είναι το πιο σημαντικό. Κατόπιν, εσείς αναφέρεστε σε μία πύλη. Φαντάζομαι ότι θα είναι δημόσια αυτή η πύλη. Πρέπει να το διευκρινίσετε κατά πώς είναι δημόσια ή ιδιωτική η πύλη όπου οι πολίτες ε, αποκτούν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές ταινίε και σε άλλες ε, εκδηλώσεις όπως είναι κοντσέρτα και θέατρο. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κατανοώ το να υπάρχει όπως την τηλεόραση, η συνδρομητική τηλεόραση, η δωρεάν ταινίε. Αλλά τώρα αυτή την πύλη, πώς ακριβώς η πύλη αυτή θα ε, συνδεθεί με τη δική μας την τηλεόραση, την τηλεόραση χωρίς σύνορα και πώς αυτή θα προσφέρει ε, την πρόσβαση σε κονσέρτα, σε συμφωνικές ορχήστρες, σε, σε θέατρα, αυτά δεν τα καταλαβαίνω και για να έχει κανείς ε, και η μία πύλη που θα δίνει την πρόσβαση σε ταινίες πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα ε, του copyright των πνευματικών δικαιωμάτων και τα παρεμφερή. Και μετά μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή. Μετά την τελευταία σύστηση που είχαμε, ακριβώς ε, η Ευρωπαϊκή είναι η δημόσια βιβλιοθήκη αυτών όλων των πολιτιστικών αγαθών, αν το καταφέρουμε βέβαια και τηρώντας όλους τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Εσείς τώρα λέτε ότι αυτό δεν θα είναι ε, ανταγωνισμός στην Google ή στην Books, αλλά θα είναι προσθήκη, που σημαίνει ότι ακόμα και αν το θέλαμε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνιστέ στην Google. Η Google είναι πολύ πιο προχωρημένη και βλέπετε κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση τι κέρδη προσπορίστηκαν αυτοί. Άρα το θέμα δεν είναι το να θέλουμε ή να μην θέλουμε, δεν μπορούμε και να θέλουμε. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι μας, ότι πρόκειται για, ένα, για μια συμπληρωματική δημόσια προσφορά, η οποία ε, δίνει τη δυνατότητα μιας ποιοτικής προσφοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λούκεγκάρτ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ε, με την ομιλία σας σε γενικές γραμμές ε, συμφωνώ με την εκθεσή σας και θα ήθελα επίσης να μπορέσω και εγώ να προσθέσω κάτι. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια, κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σημεία που θέλω να θίξω για την έκθεσή σας. Νομίζω όλοι που βρισκόμαστε εδώ συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, δίκτυο, διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Και υπάρχει και το θέμα πώς ακριβώς αυτό τελικά θα το πετύχουμε. Πώς θα ε, πετύχουμε τη στρατηγική μας και όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος ε, Μπαρόζο είπε στο έγγραφό του ε, για τη στρατηγική του 2020 ότι θέλει να εξετάσει και το θέμα των οπτικών ινών ως ένα στοιχείο της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το δίκτυο. Βεβαίως, ο ιδιωτικός ε, τομέας ε, μπορεί κανείς ε, να σκεφτεί ότι θα μεριμνήσει μόνος του. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι η αγορά είναι εκείνη που θα πρέπει να ορίσει τι, ποιες είναι οι εξελίξεις που επικρατούν. Κομισιόν έχει καταθέσει προτάσεις για κρατικές ενισχύσεις σε, κάποιους ε, φορείς και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να αναφέρεται στην έκθεσή σας. Εγώ είμαι υπέρ των ε, ΣΔΙΤ που είναι πάρα πολύ δημοφιλή και νομίζω ότι αποτελούν μια λύση αν θέλει κανείς να διαδώσει την τεχνολογία. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική αγορά, αλλά και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν θέλουμε να έχουμε υψηλότερες ταχύτητες, πρέπει να υπάρχει και ένα είδος παρέμβασης από το κράτος. Ε, ίσως και αυτό μπορείτε να το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Κατόπιν, όσον αφορά τώρα τους ε, νέους, συμφωνώ το πρόβλημα είναι με τους νέους ε, και στην έκθεσή μας νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς ε, οι ηλεκτρονικές, τα δεξιότητες μπορούν να διαδοθούν και σε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν προσόντα όπως είναι οι ηλικιωμένοι ή αυτοί που ζουν στις ε, περιφέρειες οι νέοι σε τελική ανάλυση έτσι καλώς τα καταφέρνουν βεβαίως και αυτοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αλλά θεωρώ ότι πρέπει πάνω απ' όλα να προβάλλουμε εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που βρίσκεται λίγο πιο πίσω στα στατιστικά μας δεδομένα. Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, και αυτό το ε, δευτερογενές ε, όφελος που θα προκύψει και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. αυτή η όλη διαδικασία είναι ένα τμήμα της στρατηγικής 2020. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται τις ε, εμπορικές ανταλλαγές μέσα από το διαδίκτυο και το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για πειρατεία και πνευματικά δικαιώματα, παρότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα πρέπει ως Επιτροπή να πούμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη θέση επ' αυτού και οφείλουμε να υπογραμμίσουμε το δικαίωμα ε, κάποιων καλλιτεχνών ε, το εισόδημά τους ε, να καλύπτεται. Τέλος, όλους μας μας ενδιαφέρει το διαδίκτυο αλλά δεν μπορούμε αυτό να το συζητάμε ως ε, ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρέπει να το εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος κυρία Κάμα Έμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω ότι είμαι ευγνώμων στο συνάδελφο κύριο Ήβαν, ο οποίος ε, ξεκινώντας είπε ότι η έκθεση αυτή θέλει να προβάλλει περισσότερο τους καταναλωτές. Εγώ το σχέδιο της ε, Κομισιόν το βρίσκω λιγάκι φτωχό, γιατί παρότι βεβαίως ε, η ηλεκτρονική ατζέντα θα φέρει κάποια οικονομικά ωφέλη και σωστά προβάλλεται αυτό. Δεν πρέπει όμως να παρούμε, παραμελούμε και την κοινωνική πτυχή της ηλεκτρονικής ατζέντα να το κάνουμε καλύτερα από ό,τι το κάνουμε μέχρι τώρα και ίσως αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε στην εκθεσή μας. Στην πρόταση κομισιών λείπουν και έννοιες όπου την προηγούμενη εβδομάδα Προσπαθήσαμε στην έκθεση της κυρίας ε, Γκρός ε, να αποκτήσουμε τέτοιου είδους έννοιες όπως ε, ουδετερότητα του δικτύου ή διαλειτουργικότητα των δικτύων. Όλα αυτά πραγματικά έχουν υπεραξία για τους καταναλωτές. Και αυτά είναι τομείς όπου ως Κοινοβούλιο οφείλουμε να λάβουμε σαφή θέση. Θεωρώ εξάλλου ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ηλεκτρονική συμπερίληψη ε, δεν είναι το μόνο που έχει να κάνει με την αρμοδιότητα των μέσων ενημέρωσης. Η διασύνδεση παιδείας και φτώχειας έχει ήδη αναφερθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε τελικά το όλο και διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα σε όσους έχουν εξοικειωθεί με τεχνολογία και στους υπόλοιπους, πώς θα μπορέσουμε να το συρρυκνώσουμε. Και αυτό δεν είναι στη τελική ανάλυση μόνο θέμα προσόντων, αλλά και δυνατότητων πρόσβασης σε αυτές τις νέες δυνατότητες. Θέλω λοιπόν ότι στην Ευρώπη πρέπει να βρούμε μία απάντηση η οποία θα εμποδίσει τη διεύρυνση του χάσματος και γιατί όχι να προσπαθήσουμε και να κλείσουμε και το χάσμα. Και ένα άλλο το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα και νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Επιτροπή Πολιτισμού είναι όλος αυτός ο τομέας ε, της διασφάλισης, της πληροφορίας ε, και της ε, πολιτισμικής πολυμορφίας. Γιατί όταν μιλάμε για την ηλεκτρονική ατζέντα, πολύ συχνά μιλάμε για θέματα που εμφανίζονται στο τηλεπικοινωνιακό πακέτο, δηλαδή για την ουδετερότητα των υπηρεσιών και των τεχνολογιών. Ως Κοινοβούλιο επιτύχα σημειώσαμε μια μεγάλη επιτυχία, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες ε, εξαιρέσεις από αυτήν την ουδετερότητα, αλλά μόνο προς το κοινό καλό και για τη διασφάλιση ε, της ε, πολιτισμικής πολυμορφίας. Αυτό είναι ένα θέμα που εγώ θα ήθελα στη δική μας τη γνωμοδότηση να προβληθεί ιδιαίτερα. Αναφέρομαι βέβαια στη γνωμοδότησή μας για την ψηφιακή ατζέντα. Να μην τα βλέπουμε όλα κάτω από το πρίσμα της αλλά ακριβώ το θέμα της ελευθερίας ενημέρωσης και της ε, πολιτισμικής πληροφορίας, αυτά, με συγχωρείτε, πολιτισμικής πολυμορφίας, όλα αυτά να τα προβάλλουμε ιδιαίτερα. Ο συνάδελφος κ. Μπίσκε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να, να προβάλλω κι εγώ ένα πράγμα. Ε, νομίζω έγινε ήδη λόγος. Εγώ θέλω να φερθώ στην ε, αρμοδιότητα για θέματα ενημέρωση, στα ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές εξελίξεις. Γιατί τελικά, αν είναι αλήθεια ότι ε, τα ψηφιακά εργαλεία είναι, θα είναι η τέχνη του μέλλοντος, τότε πρέπει κανείς να πει ότι οι εξελίξεις ε, δεν είναι ικανοποιητικέ. Και θα αναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Την εποχή της τηλεόρασης υπάρχουν, υπάρχουν αναλφάβητοι σε οπτικοακουστικά μέσα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ικανοί κάμεραμεν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν φωτογραφικές μηχανές και είναι εξοικειωμένοι με το ε, επάγγελμα. Κάθε τρίτο σήμερα γυρίζει ταινίε με το δικό του το βίντεο. Γιατί δεν έχουμε λοιπόν τους καλύτερους σκηνοθέτες. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα κλειδί του μέλλοντος είναι το πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε περισσότερες ικανότητες με αυτά τα ψηφιακά μέσα. Ε, όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν εξαρτώνται απόλυτα από τη θέλησή μας και καλό είναι αυτό. Δεν είναι ανάγκη όλοι να εξαρτώνται από την βούληση των πολιτικών και της πολιτικής. Το Google είναι απαραίτητο σε όλους μας, θα παραμείνει χρήσιμο και απαραίτητο, είτε μας αρέσει είτε όχι, αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε περισσότερες ε, ικανότητες στον ψηφιακό χώρο και αυτό σε σχέση με τον πολιτισμό. Ο κύριος Σμιτ. Van egy olyan német közmondás, tisztelt elnök asszony, hogy Schuster ε, Λέμε και στα γερμανικά λέγεται αυτό, δεν θα πρέπει κανένας να παραμείνει στο επάγγελμά του, δεν θα πρέπει να τρέχει από εδώ και από εκεί. Εδώ νομίζω όμως στην Επιτροπή μας θα έπρεπε να ασχοληθούμε με θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Πώς δηλαδή αυτή η ψηφιακή ανεπανάσταση μπορεί να ωφελήσει τον πολιτισμό. Η Ευρώπη νομίζω ειστερεί εναντί των ανταγωνιστών τους, της ΙΠΑ δηλαδή και της Ιαπωνίας. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν κάποιες ιδέες, μπορούν παραδείγματος χάρη να συγκεντρώσουν σε λίγο χώρο πολυμουσική, έχουν διάφορες ιδέες, πώς μπορεί κανένας να διαβάσει ηλεκτρονικά βιβλία, Κάθε δεύτερος επιβάτης στα αεροπλάνα στην Αμερική διαβάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Αυτό είναι παραδείγματο χάρη ένα τομέα στον οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Η ευρωπαϊκή μουσική, ο ευρωπαϊκό πολιτισμό θα πρέπει να προωθηθούν μέσω των νέων αυτών τεχνολογικών δυνατοτήτων. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει, όπως σας λέω, στην πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, έχουμε ελλείψεις όσον αφορά τι αναπτύξει. Είμαστε αργοί γραφειοκράτες και στις 27 χώρες μέλη ακολουθούν 27 διαφορετικοί τρόποι. Δεν είμαστε ανταγωνιστές στο Google, προφανώς απέχουμε πόρο αυτού. Αλλά ίσως θα ήταν καλό πραγματικά να έχουμε μια πύλη που θα προωθεί τον πολιτισμό. Και να έχουμε προβλήματα ερευνητικά και ανάπτυξη στον τομέα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι άμα αρχίσουμε στους μαθητές για τα σχολεία, γυμνάσια, λύκα κλπ. Τους, τους λέμε τι θα γίνει με το, με το διαδίκτυο, θα αργήσουμε. Γιατί δεν πάνε όλοι στα σχολεία αυτά. Θα πρέπει λοιπόν εκ μιας αρχής να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές στο δημοτικό. Προσπαθήσαμε παντού στην Ευρώπη να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές. Κατ' εξαίρεση συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Σπίσκι. Θα, άμα το ακούσει κανένα στην ομάδα μου θα με σκοτώσει κύριε Σπίσκι. Έχει δίκιο όμως ο κύριος Σπίσκι γιατί αναφέρεται στην πολιτιστική πολυμορφία στο κείμενό σας δεν αναφέρεται αυτό ρητά. Εγώ θα να παρακαλέσω τον κύριο Μπίσκι να υποβάλει μια σχετική τροπολογία. Αλλιώς θα την υποβάλω εγώ ή ας την υποβάλουμε και από κοινού. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που είναι η δουλειά μας να συμβάλλουμε ε, στην ε, έκθεση μιας άλλης επιτρόπης να γνωμοδοτήσουμε δηλαδή για τα πολιτιστικά. Και το European θα πρέπει να έχει πραγματικά μία δική του υπόσταση. Να μην πούμε «Ε, είναι κάπως σαν το Google και εμείς κάπου εκεί κοντά πάμε. Όχι. Όχι. Ε, βέβαια δεν πρέπει να εφεύρουμε τα πάντα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τι έχουμε ήδη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα διατυπώσουμε τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετήσουμε κανένα πολίτη εάν του δώσουμε έτσι ευρωπαϊκές ταινίε. Το copyright που θα είναι, ποιος θα πληρώσει. Λοιπόν, ας είμαστε κάπως προσεκτικοί στη διατύπωσή μας. Ας τακτοποιήσουμε κάπως το κείμενο και ας τονίσουμε αυτό που μας διακρίνει από την Επιτροπή Ήτρε. Πολιτισμός, παιδείας. Και γι' αυτό η ιδέα σας να έχουμε ευρωπαϊκές εκστρατείες στο επίπεδο αυτό, ότι θα πρέπει να σχετίζονται και με το European. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει αυτό. Δεν θα το δεχτούν ίσως όλοι, αλλά και αυτή η προσφορά στην οποία αναφερθεί δεν θα γίνει δεκτή από όλους. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε σε αυτά που μπορούμε. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να αναδιατυπωθούν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ακρόαση με ενδιαφερόμενους ε, ε, ηθοποιούς για να βρούμε τη λύση για τα, το βίντεο του μήνα. Δεν ξέρω πώς το φανταστήκατε εσείς. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το θέμα και που θα ασχοληθούν να σας παρακαλέσω να υποβάλουν λέω τροπολογίες ούτως ώστε ακριβώς για να τονίσουμε τον πολιτιστικό και ε, εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δικής μας Επιτροπής. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι παρούσα. Παρακαλώ. Θέλετε να γνωμοδοτήσετε. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση εδώ και θεωρώ πράγματι ότι η συμβολή δική σας θα πρέπει να τονίσει αυτό που είπατε κι εσείς. Και θα ενδιαφέρομαι πολύ να ακούσαμε τις απόψεις σας. Και η Κομισιόν, βέβαια θα λάβει υπόψη αυτά που έχει να πει το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Κανένας από τους αδελφούς θέλει. Ο κύριος Ιβάν, τελευταίος, για να απαντήσει. Δεν Είχα πάρα πολύ μεγάλο χώρο για το κείμενο, όπως γνωρίζετε. Δεν μπόρεσα να βάλω τα στοιχεία που επιθυμούσα στο κείμενο. Δεύτερον, αναφερθώ στο εξή. Ε, στοχεύω κυρίως τους νέους γιατί αποτελούν το πλέον δυναμικό κοινωνικό περιβάλλον και η Ευρώπη θέλει να καταστεί σημαντικός ε, παράγοντας στη διεθνή σκηνή. Εδώ μιλάμε για όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες. Υπάρχει διάκριση, υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ε, μαθητών ε, που φοιτούν σε σχολεία στις μεγάλες πόλεις ε, και έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές σε σχέση με μαθητές που μένουν σε αγροτικές περιοχές και οι ευκαιρίες που έχουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία σε σχέση με όσους ζουν σε αστικά περιβάλλοντα διαφέρουν. Και φυσικά σε διαφορετικές ε, περιοχές της περιοχέ Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρουν ευκαιρίες. Όταν μιλώ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-government, ε, δεν αναφέρομαι μόνο στο κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά έχω κατά νου και τη διαβίου μάθηση, την επαγγελματική σύγκληση και την προσαρμογή στην αγορά εργασίας όσων ε, χάνουν τις δουλειές τους. Τώρα διανύουμε μία περίοδο όπου βλέπουμε ριζικές αλλαγές ε, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην ε, παγκόσμια οικονομία. Τώρα, όταν αναφέρθηκα στην πύλη, είχα κατά νου ε, μια δημόσια πύλη όπου θα εμπλέκονται τα κράτη-μέλη και κάθε κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει πώς θα προωθήσει το δικό του πολιτισμό ως τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού φυσικά. Όταν έκανα την ε, παρουσίασή μου δεν αναφέρθηκα στη χρήση του τεχνολογίας βίντεο κατά παραγγελία, video on demand, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των δικαιωμάτων, του copyright και του πώς θα διαχειριστούμε την πρόσβαση του ευρέσκηνου στην πύλη αυτή. Αυτό δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Ε, υπάρχουν περιορισμοί που μας δεσμεύουν. Κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει να διαχειρίζεται το δικό του ρυθμιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να ρυθμίζει με ποιο τρόπο μπορεί να παράσχει πρόσβαση ε, σε κάθε ένα Ευρωπαίο πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να συστήσουμε αυτό το πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έτσι ώστε κάθε ένας πολίτες στην Ευρώπη να συνειδητοποιεί ότι είναι τμήμα τη ευρωπαϊκής οικογένειας και ότι υπάρχει ένας κοινό πολιτισμό που μας ενώνει όλους. Σε ό,τι αφορά το ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί ΙΠΑ και Ιαπωνίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα να επανέλθω σε όσα είπα πριν. Θα πρέπει να βασιστούμε στην καινοτομία των ε, νέων γενεών που κατανοούν ε, τις νέες τεχνολογίες ε, των πληροφοριών και των επικοινωνιών και που μπορούν να συνεισφέρουν με τη δημιουργικότητά τους και την κοινοτομία τους. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε τους ανταγωνιστές μας και θα κερδίσουμε εκ νέου μια ηγετική θέση. Είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένε και η Ιαπωνία προσελκύουν ε, νέους, ε, προσφέροντας τους υποτροφίες και ίσως γι' αυτό έχουν αυξημένη ανταγωνιστικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, προωθώντας τις τεχνολογίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, Όταν προωθούνται οι τεχνολογίε αυτέ, οι Ευρωπαίοι πολίτε θα συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ύπαρξη των τεχνολογιών και θα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την ασφάλεια των πληροφοριών. Θα πρέπει να το επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και έτσι οι πολίτε θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μιλώντα γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει τη συμβατότητα με άλλα συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες σας απάντησαν, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω. Κοιτάξτε, ε, την, ε, δυστυχώς τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου, είναι καταληκτική ημερομηνία που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα πρέπει να καταθέσετε τις ε, τροπολογίες σας για να έχετε προλάβει την ημερομηνία τη Δευτέρα, 12 η ώρα, 1η Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε στις 22 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιβάν, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Πάμε στο επόμενο σημείο, διακυβέρνηση του ίντερνετ, τα επόμενα βήματα. Η επί της ουσίας είναι αρμόδια η Ήτρε και εδώ ισχύει το ίδιο. Ε, μέχρι την ε, Δευτέρα, 12 η ώρα, έχουμε ε, την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Ο Ήβο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Θα ήθελα να σας πω ότι για το θέμα αυτό έχουμε συζητήσει διεξοδικά, δεν θέλω να παναλάβω τα πάντα, απλά λιγάκι να σας επισημάνω περί τίνος ε, πρόκειται. Και ε, θα κάνω τη διαπαρατήρηση όπως ε, έγινε και στην προηγούμενη έκθεση, δηλαδή πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότησης, όμως τα περιθώρια που υπάρχουν για γνωμοδότηση είναι περιορισμένα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μας ε, συνεβούλευσαν να καταθέσουμε τις προτάσεις μας το συντομότερο δυνατόν και γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι θα μας ε, βοηθήσετε το συντομότερο δυνατόν. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για το εξής. Πρόκειται για τον έλεγχο του διαδικτύου το οποίο βρίσκεται στα χέρια επιχειρήσεων ε, κοινοφελών ε, οργανισμών ε, με τα αρχικά ICON αφορούν την διεθνή συνεργασία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ιδιωτικοί οργανισμοί που μπορούν να μπορούν να ασκήσουν έλεγχο στο διαδίκτυο. Η Κομισιόν έχει καταθέσει ένα πολύ καλό, ε, περιεκτικό κείμενο και εκεί πρόκειται για τον αυτοέλεγχο του διαδικτύου, το οποίο ε, μέχρι τώρα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, όμως το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε τρωτοί. Τρωτοί κυρίως όσον αφορά την ε, διεθνή διακυβέρνηση. Αν ε, φέρει κανείς κατά νου, παραδείγματος χάνει το τι συνέβη πέρυσι στον χρηματοπιστωτικό τομέα, νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι το κράτος ε, στον τομέα αυτό πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ενεργή όσον αφορά την, ε, ε, τον έλεγχο του ίντερνετ. Αναφέρθηκε ήδη ότι πρόκειται για γνωμοδότηση για την Επιτροπή Βιομηχανίας Δηλαδή η δική μας γνωμοδότηση δεν αφορά τεχνικά στοιχεία, αλλά αφορά τα στοιχεία εκείνα που είναι σημαντικά ε, σε σχέση με τη διδασκαλία και τον πολιτισμό. Σας είπα λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης, με συγχωρείτε. Και κατά τα άλλα ε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τη διαχείριση του διαδικτύου έχουμε τον Αμερικανικό Οργανισμό Μεταρχικά ICAN και πέρα από αυτόν υπάρχουν ε, και άλλοι κοινοφελείς οργανισμοί. Αυτό στον οποίο αναφέρομαι είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι υπόλογος μόνο στην Καλιφόρνια. Και πέρυσι συνήφθη μια νέα σύμβαση ανάμεσα στην ε, Καλιφόρνια την Πολιτεία της Καλιφόρνια και την Icon Corporation. Αυτή η συμφωνία είναι καθοριστική ε, για τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Ε, έγιναν και κάποιες βελτιώσεις. κατόπιν ακολούθησε και μία επανεξέταση μέσα από ένα review panel η επιχείρηση αυτή ε, θέλει και πρέπει να είναι πιο διαφανής ε, και να είναι περισσότερο υπόλογη, καθότι ε, έχουμε ένα ευρύτερο δίκτυο με πολλούς παίκτες. Επ' αυτού όμως θα πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα προσφέρει αυτή η Επιτροπή Αναθεώρησης. Τι είναι λοιπόν αυτό που επιδιώκουμε εμείς, τι επιδιώκει η Κομισιόν, εδώ υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιθυμούσαμε μια εσωτερική μεταρρύθμιση της ε, ΙΚΑΝ, δηλαδή επιθυμούμε την πλήρη διαφάνεια και επιθυμούμε επίσης η ΙΚΑΝ αυτή να είναι υπόλογη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους ε, διεθνείς παίκτες και όχι μόνο ε, στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Με άλλα λόγια δηλαδή, επιθυμούμε την ε, ανάληψη ευθυνών σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένα πολυμερές ε, όργανο ελέγχου ε, και θα θέλαμε να γίνουν σχετικές διαπραγματεύσεις για όλα αυτά που προανέφερα. Όπως λοιπόν σας είπα ήδη, εμπνευστήκαμε και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν θέλω τώρα να σας επαναλάβω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά όπως σας είπα, ενάυσματα πήραμε και από αυτό και το 2008, δεν έχει περάσει και πολύ καιρός έκτοτε, ε, κατατέθηκε μία πρόταση για το δεύτερο φόρουμ που έλαβε χώρα στο Rio de Τζανέιρο. Ναι, εμείς καταθέσαμε ένα ψήφισμα και στο ψήφισμα αυτό αναφέρουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ε, Παραδείγματο χάρη η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, η πολυμορφία, η προσπελασιμότητα, η ανταλλαγή γνώσης Όλα αυτά αναφέρονται στο ψήφισμα του 2008, όπως επίσης και μία σειρά άλλων πραγμάτων που εφήγησαν και αποφασίστηκαν ε, στο φόρουμ του de Janeiro. Κατά τα άλλα, θα ήθελα ε, να σας πω τι είναι εκείνο που επιθυμούμε διακαώς να αποφύγουμε. Αυτό το έχω συζητήσει με τον συνάδελφό μου που είναι ο σκιώδης εισηγητής της Επιτροπής Βιομηχανίας και νομίζω συμφωνούμε όλοι μας ε, ότι ε, όσον αφορά το τηλεπικοινωνιακό πακέτο θέλουμε την ουδετερότητα Επιθυμούμε λοιπόν να μην επανέλθει το τηλεπικοινωνικό πακέτο σε αυτή τη συζήτηση. Επ' αυτού θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι. Κατά τα άλλα, η συζήτηση για το ε, ψηφιακό περιεχόμενο και αυτή πρέπει να αποφευχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο. Υπάρχουν ε, άλλα εργαλεία, άλλες εκθέσεις, ε, αλλά εν πάση δόση, εγώ είμαι ανοιχτός για συζήτηση ή για κριτική για αυτά που σας λέω τώρα. Τώρα πάμε στη γραμμοδότηση. Είναι το έγγραφο υπαριθμών 6. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σειρά αρχών που είναι πολύ σημαντικές για μας. Δεν θέλω να τις ε, επαναλάβω. Πρόκειται για την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, πολυμορφία, πολυπλουραλισμό, σημεία 5 και 6. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει με απόλυτη σαφήνεια ότι πρέπει να ε, λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι ώστε πραγματικά ε, να καταλήξουμε σε περισσότερο υπεύθυνη και διαφανή, διαπραγματεύσει, διαπραγματεύσεις, διατλαντικές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε το ίντερνετ να είναι πραγματικά ελεύθερο και ασφαλές σε ολόκληρο τον κόσμο πριν από μερικές εβδομάδες, το έγραψα ήδη αυτό, ε, αλλά ε, αν δει κανεί τι συμβαίνει στην Κίνα, νομίζω ότι το θέμα είναι πλέον ιδιαίτερα επίκαιρο και ε, θα καταστεί όλο και περισσότερο επίκαιρο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να αποφύγουμε να ξαναβρεθούμε σε τέτοια θέση. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με την ε, παγκόσμια ε, διαχείριση του ίντερνετ ε, που ξεκινάει από την Καλιφόρνια, αλλά είμαστε ιδιαίτερα τρωτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Θα αφήσω κατά μέρο κάποια θέματα, αλλά πάω στο πρώτο τελευταίο, στο υπαριθμόν 8. Εκεί λοιπόν είναι, καθίσατε σε η σημασία πρωτοβουλειών και δράσεων υπέρ της προστασίας των ανηλίκων. Ε, το πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του ίντερνετ το γνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, θα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο. Εμάς ε, μας ενδιαφέρουν και άλλες πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά την κυβερνοεγκληματικότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια είχα να σας πω αποτελούν μία περίληψη ε, του σχεδίου της ε, γνωμοδότησης ε, και όπως σας είπα είμαστε ανοιχτοί για προτάσεις τροπολογίες οι οποίες όμως δυστυχώς πρέπει να κατατεθούν το συντομότερο δυνατόν εγώ. Ήταν πολύ πλήρη η παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω στους, ε, τους συναδέλφους να κάνουν κάποιες ε, παρατήσεις αν έχουν. Μαρία Φαντεφούτσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριο Μπέλετ ε, για αυτή την γνωμοδότηση. Έχω κάποια σχόλια που αν έχω χρόνο θα ήθελα να τα μεταφράσω σε τροπολογίε. Όμω δεν ξέρω θα προλάβω γιατί δεν ξέρω ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία. Αναφερθήκατε ε, στο ότι λάβατε ω βάση το ψήφισμα που υλοποιήσαμε το 2008 μετά το Ρίο. Όμως το 2009 είχαμε και ένα άλλο φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου στην Αίγυπτο και υπήρξαν περισσότερες πληροφορίες εκεί που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη σε ψήφισμα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να το συζητήσω αυτό με τον κύριο Μπέλετς, ό,τι αφορά το ICAN. Ε, η αλήθεια είναι ότι είπατε ότι πέρσι τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκε ε, μία ε, σύμβαση και ολοκληρώθηκε αυτό που είχε, ε, μάλλον η θητεία του ΆΙΚΑΝ ολοκληρώθηκε και τώρα βρίσκεται αυτό στα χέρια μιας επιτροπής. Πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα αυτό. Δηλαδή, ε, η θέση αυτή είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κέρδος δικό μας, γιατί αυτό έφυγε από τα χέρια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

και είπατε ότι θέλετε να εξεύρουμε ένα πιο πολυμερέ σύστημα. Όμω αυτό ενέχει κινδύνου. γιατί αν ε, ε, λάβουμε υπόψη και τη βούληση τη Κίνα, θα σημαίνει ότι και αυτή θα θέλει να συμμετάσχει, Όμω ε, αυτό δεν αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη διαχείριση του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν είναι κάπως πιο πολύπλοκο το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα δύο τελευταία σημεία, 8 και 9, που αναφέρονται στην προστασία των ενηλίκων όταν χρησιμοποιούν το ίντερνετ στο Σάρμελ Σέιχ, ήδη προέκυψαν διάφορες προτάσεις, ε, δηλαδή να, δίνονται, ε, να δίνεται υλικό έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες να μπορούν να καταρτίζονται έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να ελέγχουν την πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο αυτό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και εγώ θα ήθελα να ε, φέρω ορισμένα στοιχεία που προέκυψαν από τη συζήτηση στο Σάλμεν Σέιχ τον περασμένο Νοέμβριο. Αν προλάβω τι ημερομηνίε, θα ήθελα να υποβάλω αυτέ τι τροπολογίε. Σα ευχαριστώ. Η uh, thank you very much, Chair. Um, just... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μας ε, το σχέδιο ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπελέ είναι πάρα πολύ καλό για έναν ιδιαίτερα ευρύ τομέα και θεωρώ ότι ε, την τελευταία φορά ήμουν εδώ και είχαμε μία ε, μακρά ανταλλαγή υπόψη. Δεν χρειάζεται τώρα πάλι να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ και δύσκολο τομέα για να καλυφθεί. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι το σχέδιο αυτό πράγματι καλύπτει την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει πρόεδρο, δεν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση. Αν όχι, παρακαλώ ο Ήβο για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ τώρα. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Υπήρχε στο σαμεσέ είχε αυτό το φόρουμ διαδικτύου. Δεν ήμουν παρόν, αλλά το ευεστερό ήταν εκεί και άλλοι και αύριο θα έχουμε στο κοινοβούλιο, στο, εδώ στο εστιατόριο, ένα πρόγευμα πάνω στο θέμα, στις 8 το πρωί, ένα πρόγραμμα εργασίας. Ο Σφίνης εδώ θα είναι παρόν και θα επαναλάβει ακριβώς τι ελέγχθη όσα μας έχει. Αν ενδιαφέρεται κανένας, έχω εδώ τις, ε, τα έγγραφα του το ελέγχθη Σάικ. Είναι πολύ ελληνικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό που ανεφέρθη στο θέμα αυτό και θα περιμένω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας, θα το λάβω υπόψη μου. Αυτό που είπατε για, την πολυμερή, για το πολυμερή έλεγχο ε, είναι ενδιαφέρον, είναι βέβαια επικίνδυνο γιατί συμπεριλάμβανται και οι Κινέζοι και θα πρέπει να δούμε τι έχει να πει η Κομισιόν πάνω σε αυτό, θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον που έχουμε και να φροντίσουμε και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε καλύτερου μηχανισμού ελέγχου. Ιδίω όταν πρόκειται για θέματα τη προστασία των παιδιών θα πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε. Και εγώ έχω μια σειρά τροπολογιών που θα ήθελα να υποβάλω. Και με χαρά θα περιμένω και τι ε, τροπολογίες σχέσεις μετά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το σημείο τη μέσης διάταξη. Θα ήθελα ξανά να σα υπενθυμίσω ότι και εδώ η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, 1η, 1η Φεβρουαρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλη Νοεμβρίου, το Ελεκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια εκθέση για την ε, εκτέλεση από την Κομισιόν του Προπολογισμού του Περιορισμένου Έτους και βέβαια καλούμεθα ως Επιτροπή να ελέγξουμε κατά πόσον οι δικές μας ε, ανησυχίες καλύφθησαν και τα χρήματα που διαθέσαμε ε, διαπαντήθηκαν σωστά ή κατά πόσον τα χρήματα αυτά πήγαν αλλού, όχι εκεί που θέλαμε, για να το πω έτσι κάπως χοντρά. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια τώρα να μας εξηγήσει. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πάκ, αγαπητοί συνάδελφοι πάλι πρόκειται για το θέμα της απαλλαγής για την εκτέλεση του προπολογισμού 2008. Για το τμήμα της ε, εκτελεστικής επιτροπής και των εκτελεστικών υπηρεσιών. Από σκοπιάς μου δεν έχουμε τίποτα το δραματικό να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες προτάσεις. Θα θέλαμε, μια που πρόκειται τώρα για την μεσοπρόθεσμη θεώρηση των πολιτών προβλέψεων, να εξετάσουμε ποιες ήταν οι δομές ε, για την εφαρμογή και τη διαχείριση, για την εκτέλεση μάλλον του προπολογισμού και τη διαχείρισή του. Ιδίως θα πρέπει να δούμε πώς, κατά πόσο ήταν ικανοποιημένοι οι πελάτες. Η δική μας δηλαδή πελατεία που συμμετείχε εδώ πέτυχε αυτό που ήθελε ή δεν το πέτυχε και η τελευταία αναλύση ποιες είναι οι εμπειρίες των Ευρωπαίων πολιτών που υποβάλλουν αιτήσει όσον αφορά τον προπολογισμό αυτό και κατά πόσο συμβάλλει στην αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα πράγματα είναι εύκολα, δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτή είναι μια εμπειρία που έχω εγώ συχνά. Όταν υπάρχουν εκεί προβλήματα, υπάρχει πραγματικά έλλειψη της ικανοποίησης του πελάτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και θα ήθελα να τονίσω ότι το 70% των πόρων των πολιετών προγραμμάτων ε, εκτελούνται από εθνικές υπηρεσίες. Έχουν λοιπόν έντονη ευθύνη και γι' αυτό οι δικέ μας γνώσεις για το τι κάνουν οι εθνικές υπηρεσίες τα 27 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί εμεί θα πρέπει μετά να κρίνουμε κατά πόσον εκτελούνται πραγματικά τα πολιτικά μας προγράμματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχονται τα πράγματα ενεργά και θα πρέπει να ξέρουμε, αν θέλουμε να υπάρχει τέτοιο θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί κυρώσεων, αν τα πράγματα δεν πάνε σωστά. Και η πρόταση είναι, εάν υπάρχουν πραγματικά αδύναμα σημεία, να διακόψουμε τις πληρωμές, καλώντας να βελτιωθεί η διαχείριση, για να μην υπάρχουν προβλήματα για τους δικαιούχους. θα πρέπει να δούμε, όπως λέγεται ο στόχος είναι η μεταβίβαση των γνώσεων για την Ευρώπη και να τονίσουμε ότι υπάρχει αυτός ο σημαντικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και ότι θα πρέπει η εργασία στον τομέα της ε, πολιτικής επικοινωνίας να είναι τέτοιος, ωστόσο ώστε πραγματικά η κοινωνία των πολιτών να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, πρέπει εμείς να δράσουμε, αλλά θα πρέπει βέβαια να έχουμε και τους άλλους που να συνεργάζονται μαζί μας. Και θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων εδώ και του τι γίνεται επιτόπου στα κράτη-μέλη, στους δικαιούχους. Και τέλος, όσον αφορά την ε, ανάγκη διάθεση πραγματικών πόρων για τα ε, κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά ενεργό πολιτική επικοινωνία. Να φροντίζουμε το ώστε να είναι γνωστό ότι είναι καλό αυτό που κάνουμε. Και θα πρέπει να βρούμε τις σωστές ε, μεθόδους για να το πετύχουμε. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαθέσουμε όχι μόνο εμεί πόρου, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει σημαντικά να διαθέσουν άλλους πόρου. Ευχαριστώ. Προέδρο, ευχαριστώ. Χέλγα, τι έχουν ζήσει λόγο, ο κύριο Μάτιν και ο κύριο Μπέλετ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε αγαπητοί συνάδελφε κυρία Τρούπελ. Μόνο μία ερώτηση θα μου επιτρέψετε. Λίγα, αυτά τα διοικητικά έξοδα, τις διοικητικές δαπάνες, εκεί ε, μήπως ε, μπορείτε να προτείνετε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη λεπτομέρεια κυρίως και εν πάση περιπτώσει αν δεν το κάνετε εσείς ε, θα δεχθείτε να καταθέσουμε εμείς σε μια τροπολογία ή αν θέλετε θα στηρίξετε μια δική μας πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση ο Ήβο και εγώ ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ ε, πράγματι η διαφάνεια σημαντική και ο ρόλος της κοινωνίας και η φιλικότητα προς ε, τον καταναλωτή. Είναι καλή λοιπόν αυτή η πρόταση σχετικά με τις ερωτήσεις προς τον καταναλωτή. Βεβαίως ε, θεωρώ ότι όλα μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, κυρίως όταν πρόκειται για διαφάνεια. Και μπορούμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε ε, κάποιες αποφάσεις ε, να χρησιμοποιούνται καλύτερα σε σχέση με τις ενισχύσεις. Και επιτρέψτε μου και μία άλλη ε, παρατήρηση. Όταν πρόκειται για επαφές με οργανισμούς και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται για τον πολιτισμό και όταν πρόκειται για εθνικούς φορείς, νομίζω ότι είναι σημαντικό η Κομισιό να καθορίζει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να τις ακολουθεί. Βέβαια, επανειλημμένα έχει ασκηθεί κριτική ότι εδώ είμαστε ιδιαίτερα τυπολάτρεις, ε, ότι οι αυστηροί αυτοί κανόνες δεν ταυτίζονται πλήρως ε, με την πράξη. Ως εκ τούτου η Κομισιόν ίσως θα πρέπει να δείχνει μια μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως όσον αφορά την προσαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών. Και κυρία εισηγήτρια θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο ε, που το έχω πάρει από τη γνωμοδότηση του 2007. Εκεί πρόκειται για κανόνες και αρχές που αφορούν στο κέρδος, ότι δεν πρέπει να ε, προκύπτει κέρδος. Ε, νομίζω λοιπόν αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες για να ε, μπορούν να χορηγηθούν ε, και ε, ευνοϊκές, να υπάρξει ευνοϊκή μεταρρύθμιση χωρίς να φοβάται κανείς ότι με τον τρόπο αυτό μέσα από τη συγχρηματοδότηση θα λάβει λιγότερα κονδύλια. Αυτό αποφασίστηκε το 2007. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και εφόσον αυτό ισχύει τότε μπορούμε και εμείς να το υιοθετήσουμε. Ο συνάδελφος Ιβαν έχει το λόγο. Εγώ υποστηρίζω 100% την κυρία Τρίπελ, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται διαφάνεια, όχι μόνο όταν μιλάμε για την αξιολόγηση ε, των project, αλλά χρειαζόμαστε και 100% διαφάνεια στη διαδικασία ελέγχου και εφαρμογή. Και όταν ελέγχουμε με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των προγραμμάτων από τις εθνικές υπηρεσίες, τότε δεν θα πρέπει μόνο να βλέπουμε αν υπάρχει ικανοποίηση των δικαιούχων, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις διαδικασίες συνέχισης, follow-up, όταν δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς ε, τα κονδύλια αυτά κάνουν την ποιοτική διαφορά στον τομέα που χρησιμοποιήθηκαν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πόσο δικαιούχος ε, μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δεν ε, θα έπρεπε να έχουμε μία βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, αλλά μία μεσοπρόθεσμη, ίσως και, και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τα κονδύλια αυτά. Θα πρέπει να αξιολογούμε τα αποτελέσματα για μια πιο μακρόχρονη περίοδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νάουτς από την Επιτροπή, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μπορώ να σχολιάσω τα δύο πρώτα σημεία της ε, γνωμοδότησης και νομίζω ότι ο συνάδελφος θα αναφερθεί σε συμμετρία και 4 για την ανακοίνωση της ΚΑΜΑΔΑΛΤΑ. Τώρα, το πρώτο θέμα που αφορά την αξιολόγηση. Η ενδιάμεση αξιολόγηση ήδη έχει ξεκινήσει και συμπεριλαμβάνονται στι αξιολογήσει αυτέ ερωτήσει για τη φιλικότητα προ το χρήστη, τη διαχείριση του συστήματο και πώ λειτουργούν όλα αυτά, αλλά και για το, τι μακροπρόθεσμε συνέπειε τη της χρήσης των κονδυλίων. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν τα έχουμε θίξει. Υπάρχει και έχει προβλεφθεί και μία ε, δημοσκόπηση, μια έρευνα στους δικαιούχους και θα καλυφθεί και η πτυχή της ικανοποίησης των πελατών σε αυτή τη μελέτη. Έτσι λοιπόν να συνεχίζονται αυτές οι δραστηριότητε, Βέβαια θα χρειαστεί ένας ακόμη χρόνος πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα, στο σημείο 2 καλωσορίζουμε τη διατύπωση ε, που αναφέρεται στην καθοδήγηση που δίνεται στις εθνικές αρχές, όπως αναφέρθηκε και από το ελεκτικό συνέδριο. Επίσης αναφέρεστε στη δουλειά που κάνουμε για την παρακολούθηση και την εποπτεία και για, στην αυστηρή γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε πολλές φορές κάνοντας κάποιες περικοπές ε, κονδυλίων για τις εθνικές υπηρεσίες. Σε μια περίπτωση το πράξαμε ήδη Λέγεται και στην γνωμοδότηση προσπαθούμε πάντοτε να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες ε, επί των δικαιούχων. Τώρα, για να καλύψω κάποια από τα υπόλοιπα σχόλια, Θα δούμε και τις αξιολογήσεις ε, που αφορούν τα διοικητικά προγράμματα, μάλλον τα προγράμματα διοικητικού κόστους. Και ε, να αναφερθώ στο όσο υπόθηκαν τον κύριο Μπέλετ, για τους ε, κανόνες ελέγχου των εθνικών υπηρεσιών και των εθνικών αρχών. Πολλές φορές ε, θεωρείται ότι είναι πολύ λεπτομερής ε, ή πολύ αυστηρή. Το γνωρίζουμε, τη γνωρίζουμε αυτή την κριτική. Είναι δύσκολο να εξεύρουμε την ισορροπία. Συνεχώς προσπαθούμε να απλοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο, ενώ διατηρούμε και το απαραίτητο επίπεδο εποπτείας και ελέγχου. Βέβαια με τις ε, μικρότερες υπηρεσίες ε, κατανοούμε ότι το άχθος μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με το άχθος ε, επί των μεγαλύτερων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος για μια υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κερδοφορίας, το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν γίνονται κάποια βήματα στην ε, αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που θα κατατεθεί αργότερα φέτος προκειμένου να δοθεί εκεί μεγαλύτερη ευελιξία. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η αρχή ότι οι επιδοτήσεις δεν οδηγούν άμεσα σε κέρδος, αλλά ίσως μπορεί να ε, τεθεί δυνατότητα δημιουργίας κάποιου αποθεματικού σύντοχρονου. χρόνο. Και φυσικά στην αξιολόγηση θα λάβουμε και το θέμα της αξιολόγησης των κονδύλων. Παρακαλώ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριος Γιώνα. No problem. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είστε στο τέλο τη συνεδρίας. Στι παραγράφου 3 και 4 καλωσορίζουμε τι συστάσεις σα. Εδώ βασικά αναφερόμαστε στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη μέσω των συμπράξεων. Ναι, φυσικά θέλουμε να σκεφτούμε περισσότερο επί των διαθεσμικών διοργανικών προτεραιοτήτων. Μην ξεχνάτε ότι το 2009 ήταν το πρώτο έτος που είχαμε ε, τέτοιες διοργανικές ε, ε, προτεραιότητες. Δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συμπράξεις διαχείρισης όχι να το περιορίσουμε στο δημοσιονομικό κονδύλι εκεί, αλλά να ξεκινήσουμε και ένα πολιτικό διάλογο με τα κράτη-μέλη για το πώς θα ε, μπλέκεται η Ευρώπη σε κάθε μεμονωμένο κράτο μέλο και φυσικά στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε την τελευταία παράγραφο τη στασή σα ε, που απευθύνεται τα μάλλα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπληρώσουν τι δικέ μα δραστηριότητε και με χρηματοδότηση από τη δική του πλευρά. Αυτό φυσικά θα το αναφέρουμε και στα κρατημέλη, δηλαδή θα πούμε ότι δεν είναι μόνο η Κομισιόν, αλλά και το Κοινοβούλιο θέλει να συνεισφέρετε κι εσείς. Και ελπίζουμε ότι θα το κάνουν. Συνολικά, συμφωνούμε πάρα πολύ με τα όσα έχετε γράψει σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Uh, ε, πρόεδρος, το μέλλον θα είσαστε αρμόδιος για αυτά τα θέματα ή θα σας τα πάρει η κυρία Ρέντινγκ και θα πάει η δουλειά σας προς τα εκεί, προς την κυρία Ρέντινγκ. Ε, η δουλειά μας θα πάει στην κυρία Ρέντινγκ, αλλά όχι εμείς, που σημαίνει ότι εγώ... Και η δουλειά μας και εμείς θα πάμε, με σχόλια στην κυρία Ρέντινγκ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τα σχόλια των συναδέλφων από την Κομισιόν. Χαίρομαι που θα υποβάλλετε τροπολογίες και έτσι όλα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και θα μπορώ και εγώ να δω τι ακριβώς επιθυμείτε. Να κάνω μία παρατήρηση, γιατί το έθιξε το θέμα ο κύριος Μπέλετ. Πρόκειται για την διαμάχη που υπάρχει σχετικά με τα οικονομικά, τη ρύθμιση των οικονομικών καλούμεθα να είμαστε πάρα πολύ λεπτομερεί ε, για να μην δημιουργούνται σκάνδαλα. Από την άλλη, βέβαια, μα λένε όχι υπερβολικέ ρυθμίσει, κυρίω στα μικρά προγράμματα, ε, γιατί εκεί του δυσκολεύουμε τη ζωή. Έτσι λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια τη προηγούμενη θητεία διαπραγματευθήκαμε αλλαγέ και είδαμε πόσο δύσκολο είναι οι τρει ε, θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωση να καταλήξουν σε μία λύση. Πάντω το βλέπω το πρόβλημα και ελπίζω με την υποστήριξη κάποιων συναδέλφων που ασχολούνται με το θέμα ε, να μπορέσουμε να βρούμε μία σωστή αλλά όχι λάθος ελάφρυνση των διαδικασιών. Πρόεδρος, ε, υπάρχει αυτή η παραδοσιακή συμφωνία που αφορά στα οικονομικά. Βέβαια, αυτή είναι μόνο δύο θητείες, έχει διάρκεια ζωής δύο θητείες. Παλαιότερα δεν συνέβαινε αυτό και αυτή η υπερβολική γραφειοκρατία για μικρές επιχειρήσεις που καλούνται να συμπληρώσουν χιλιάδε χαρτιά για να πάρουν στο τέλος 500 ευρώ, ε, αυτό είναι μάλλον υπερβολή. Δεν θα πρέπει λοιπόν ευθύ εξ αρχή να θεωρεί κανεί ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να εξαπατήσουν και δεν θα πρέπει όλε οι ΜΚΟ να εμφανίζονται ή να θεωρούνται ότι είναι απαταιώνε. Αλλά ξέρετε, γίνεται από την άλλη πλευρά και η Κομισιόν εκείνη φοβάται ότι θα κληθεί εκείνη να το λύσει το θέμα. Κάπου στη μέση είμαστε εμεί. Πάντω, θεωρώ ότι για μικρότερα ποσά ε, θα πρέπει να αναζητηθεί λύση ας πούμε αυτή που κάναμε ε, στις συνεργασίες ε, με τις πόλεις. Μετά από πίεση ε, των κοινοβουλίων απλουστέθηκαν τα πράγματα. Τώρα σε προγράμματα όπως το κομμένιους ή τα προγράμματα των νέων τα ποσά δεν είναι τα ίδια όπως αυτά στα ναυπηγεία στο Ρόστοκ άλλο ήταν άλλο και άλλο και ελπίζω να κυριαρχήσει η λογική. Πάμε στο ροστοκ αλλο ηταν αλλο το αλλο και ελπιζω σημείο τη σημερινή διάταξη που σημαίνει λύεται αυτή και σας παρακαλώ αύριο να είστε εδώ στις 3 και παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα οι συνάδελφοι συντονιστές. Και αν αρχίσουμε γρήγορα θα τελειώσουμε και γρήγορα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση της κυρίας Τρούπελ. Δεν υπάρχουν και παραπλές νομίζω. 29 Ιανουαρίου, 12 η ώρα. So, ich beende die Sitzung nochmal ordentlich. Jetzt bitte die Koordinatoren jetzt ganz schnell dazu. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα να μείνουν μόνοι οι μόνοι συντονιστές για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το τελευταίο σημείο